Good morning, Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ε, παρακαλώ καθίστε. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με την υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης. Υπάρχουν προτάσεις, αντιρρήσεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Όχι. Οπότε ε, μπορούμε να υιοθετήσουμε το προσχέδιο της ημερήσιας διάταξης ε, και τώρα περνάμε στην έγκριση των πρακτικών της 22ης και 23 Νοεμβρίου καθώς επίσης και 7 και 14 Δεκεμβρίου. Ε, τα πρακτικά είναι, βρίσκονται online διαθέσιμα και προτείνω ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας θα εγκριθούν. Ε, το επόμενο θέμα αφορά ανακοινώσει Προέδρου. Ε, εντάχει να σας ενημερώσω πρώτα απ' όλα στις 22 Ιανουαρίου την Δευτέρα Είχαμε μια συνάντηση της ε, ΚΟΣΑΚ, ε, της ε, Επιτροπής των Υπευθύνων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συνάντηση αυτή ήταν στο πλαίσιο, έγινε στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας. Έλαβε χώρα στην Σόφια. Προσκλήθηκα να συμμετάσχω μαζί με τον κύριο Τίμερμαντ, τον Αντιπρόεδρο και ενημέρωσα τα μέλη της ε, ΚΟΣΑΚ για το έργο της Επιτροπής ΡΕΓΙ. Το βασικό θέμα ε, της συνάντησης αφορούσε το μέλλον της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, και επικεντρώθηκα στο γεγονός ότι όλες οι γνωμοδοτήσεις μας, οι εκθέσεις μας αποτελούν μια προετοιμασία για το μέλλον της Ευρώπης και συγκεκριμένα της πολιτικής συνοχής για την Ευρώπη. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι δέχθηκαν με ευχαρίστηση την, ε, θετικά την ε, παρουσίασή μου. Ήταν μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης που αποτέλεσε, αυτό είναι και το δεύτερο κομμάτι της ανακοίνωσής μου, ο κύριος Τίμερμαντς ανακοίνωσε ε, ο, το, την έναρξη του έργου ε, της ομάδας εργασίας για την επικουρικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί από τον ε, πρόεδρο Γιούνκερ. Αρχικά η όλη ιδέα ήταν να συμπεριληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτήν την ομάδα. Σήμερα όμως έχουμε μια ομάδα εκπροσώπων από τα Εθνικά Κοινοβούλια τα οποία έχουν οριστεί από την ΚΟΣΑΚ καθώς επίσης ε, και τρία ε, μέλη της Επιτροπής των ε, Περιφερειών. Αρχικά η πρόταση ήταν να συμπεριληφθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο όμως τελικά δεν συμμετέχει σε αυτήν την ομάδα. Έτσι έχει η κατάσταση. και η όλη ιδέα είναι η συγκεκριμένη ομάδα να συζητήσει και να παρουσιάσει προτάσεις σχετικά με το μέλλον ε, της επικουρικότητας κάνοντας περισσότερα με λιγότερους πόρους. Αυτή είναι όλη η ιδέα. Το τρίτο θέμα που θέλω να ανακοινώσω αφορά ε, την, ε, ε, το σχέδιο πρότασης σχετικά με την αποδοτικότητα. θα το συζητήσουμε αυτό και θα υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε τοπολογίες. Ε, περιμένω τους εκπροσώπους από το ΕΠΠ να ε, εγείρουν ερωτήματα πάνω σε αυτό ε, και στη συνέχεια θα το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των συντονιστών. Σας καλώ όλους λοιπόν να παρευρεθείτε σε περίπτωση που έχετε κάποιες προτάσεις. Και τέλος η τέταρτη ανακοίνωση θα είναι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ε, σήμερα μετά την ε, συνάντηση θα έχουμε μια εκδήλωση για την ε, νέα χρονιά σας. Ευχαριστώ πολύ. Σχόλια, ερωτήματα. Όχι. Οπότε λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στα βασικά θεμεία της ημερήσιας διάταξής μας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ε, με την έκθεση την οποία ε, προετοιμάζει ο κύριος Βον που αφορά τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Βόρεια Ιρλανδία. Πέρσι το φθινόπωρο αποφασίσαμε να υποβάλουμε μια εκτελεστική πράξη σχετικά με, την, ε, με τις συνέπειες ε, που θα υπάρχουν για τη Βόρεια ε, Ιρλανδία. Η έκθεση αυτή θα συνεισφέρει στο έργο της Επιτροπής σχετικά με τη, σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής συνοχής και επίσης θα μας βοηθήσει στο να σχεδιάσουμε την επόμενη γενιά της πολιτικής μας. Επίσης, ε, εκφράζει και τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας όσον αφορά την αποχώρηση ε, της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συνέπειες που θα έχει αυτό για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βόν για να ε, παρουσιάσει ε, το σχέδιο έκθεσης ε, και στην συνέχεια θα σας παρουσιάσω το σχέδιο που είπα, το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου. Ε, δυστυχώς πάσχω από ανθρώπινη γρήπη. Είμαι πολύ καροποιημένο που συντάσσω την έκθεση και πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, σε σχέση με τον αντίκτυπο πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν πρόκειται να γράψουμε μια νέα έκθεση για τον Brexit, απλώ ε, θέλουμε να επικεντρωθούμε στα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ειρηνευτικό πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη της Βορειάς Ιρλανδίας ε, και την ανάκαμψή της μετά από δεκαετίες ε, πολέμου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρέχει οικονομική υποστήριξη από το 1989 για την ειρηνευτική διαδικασία, το PIS 1, 95-99, το PIS 2, 99-2006, το PIS 3, 2007-2013 και είχαμε μία συνεισφορά της τάξης των 9,3 δισεκατομμυρίων λιρών. Τώρα έχουμε το τέταρτο πρόγραμμα ειρήνης 2014-2020 με συνολική αξία 270 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 229 εκατομμύρια, το 85% έχει προέρθει από το ΕΤΠΑ. Ξέρετε ότι το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει διδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση του προγράμματος. Αυτό που θα ήθελα να κάνω τώρα είναι να σας δώσω κάποια πρακτικά παραδείγματα των ε, προγραμμάτων που λαμβάνουν ε, χώρα. Οι συνάδελφοι βέβαια εδώ γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια παραδείγματα που μας δείχνουν τον αντίκτυπο επιτόπου. Ένα παράδειγμα είχε να κάνει με την συνεργασία του project της συνεργασίας Working Together. Ε, έχουμε ε, στην συνοριακή περιοχή 12 project στον τομέα της υγείας και προωθούν την υγεία και την ισότητα σε πιο αγροτικές περιοχές. Πάνω από 50.000 ασθενείς ε, έχουν επωφεληθεί από τις υπηρεσίες ε, του προγράμματος αυτού. Ένα δεύτερο παράδειγμα έχει να κάνει ε, με ένα πρόγραμμα που λέγεται πίσω στο μέλλον και Πρόκειται για μια οργάνωση διασυνοριακή που θέλει να βοηθήσει τους νέους να ενταχθούν και να συμμετέχουν στην ειρηνευτική διαδικασία Πιστεύω λοιπόν, ε, Πρόεδρε, ότι από αυτά τα δύο παραδείγματα μπορούμε να πούμε ότι το πρόγραμμα της ειρήνης έχει κάνει τεράστια διαφορά και στις ε, δύο κοινότητες και μάλιστα θα ήθελαν κάποιοι να συνεχιστεί και μετά το 2019. Για την έκθεσή μας ε, τώρα, εγώ έχω θέσει τρία ερωτήματα στον εαυτό μου που νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσει η έκθεση. Ίσως συνάδελφοι να προσθέσουν και άλλα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε στην ε, έκθεση πώς ε, η χρηματοδότηση έχει βοηθήσει την ειρηνή, τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και τη συνοχή. Θα πρέπει να δούμε πώς έχουν χρησιμοποιηθεί σε συντονισμό τα κονδύλια με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, να δούμε σε ποιο βαθμό τα προγράμματα ε, ουσιαστικά καθοδηγούνται από την κοινότητα και πόσο επιτυχή ήταν. Και όπως είπατε εισαγωγικά κι εσείς, ε, Εμεί θέτοντα αυτέ τι ερωτήσει μπορούμε να μάθουμε ευρύτερα διδάγματα που θα είναι χρήσιμα για το μέλλον τη πολιτική συνοχή όταν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο μέλλον για τα επόμενα βήματα. Η πρόταση είναι να έχουμε μια διερευνητική αποστολή, πιθανότατα το Μάρτιο φέτος και φυσικά ανυπομονώ να ελοπιθεί η αποστολή αυτή και να συμπεριλάβω τα πορίσματα στην έκθεση και περιμένω και τις συνεισφορές των άλλων συναδέλφων σήμερα. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει η συζήτηση. And, uh, Mr. Με τους σκιώδεις ηγητές. Ας αρχίσουμε τον κύριο Φλακ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως εκπρόσωπος ε, του κόμματος ε, των συντηρητικών από τη Βρετανία ε, στην Επιτροπή μας πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Στο σύνολό του το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός συνεισφορέας. Αλλά η Βόρεια Ιρλανδία είναι καθαρός δικαιούχος των περιφερειακών ταμείων και έχει μεγάλη επίπτωση χρηματοδότηση. Εκεί βλέπουμε ποιες περιφέρειες πρέπει να βελτιωθούν. Να σας αναφέρω μερικά στοιχεία ενδεικτικά και να τα τονίσω. Πρώτον, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η Βόρεια Ιρλανδία ως μεταβατική περίοδο θα πρέπει, ε, ε, περιφέρεια μάλλον, θα πρέπει να έχει μια συνολική προσέγγιση ε, οικονομικά, και γενικότερα 835 έχουμε από το PDP ε, αλλά ε, χρειάστηκε αυτό να αντληθεί από διάφορες πηγές και διάφορα κονδύλια. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι προτεραιότητες και με επιτυχία ε, να δράσουμε για να έχουμε αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν τα κονδύλια πραγματικά πηγαίνουν εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Δηλαδή σε τοπικό επίπεδο να υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι. Και τέλος θα ήταν δύσκολο αυτή τη στιγμή να ε, τα δούμε όλα αυτά χωρίς να αναφερθούμε στο μεγάλο ταμπού που είναι το Brexit. Η ομάδα των συντηρητικών θεωρεί ότι δεν έχει καταφέρει συγκεκριμένη έκθεση να συνδυάσει τον αντίκτυπο των περιφερειακών ταμείων για τη Βόρεια Ιρλανδία με τον αντίκτυπο του Brexit για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω συνάδελφοι ότι δεν πρέπει να θίγουμε τα κακό κείμενα εκτός της δικής μας αρμοδιότητας αλλά ο τίτλος της έκθεσης είναι πάρα πολύ ενδεικτικός. Ε, είναι ο ε, αντίκτυπος πολιτικής συνοχής και όχι μια εκτίμηση για το μέλλον. Τι θα γίνει όμως με τη μελλοντική ε, πολιτική συνοχή στη Βόρεια Ελλάδα μετά το Brexit. Δεν μπορούμε να αποφεύγουμε τη συζήτηση αυτή. Το ξέρω ότι είναι έκθεση πρωτοβουλίας. Υπάρχει μια κοινή έκθεση που συμφώνησαν τα δύο μέρη, η Μεγάλη Βρετανία και ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τέλη του έτους θα ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις του και δύο πλευρές μέχρι το 2020 από το σημερινό PDP για την ειρήνη και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Στα διαρθωτικά ταμεία βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθεί να συμμετέχει μέχρι εκείνη την ε, ημερομηνία πέραν αυτής της πληροφόρηση που ακόμα εκκρεμεί ε, βάσει ε, της αρχής ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα, η Επιτροπή ε, Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης δεν θα πρέπει να εκφέρει γνώμη. Και η ομάδα μας είναι στεναρά υπέρ αυτής της άποψης και θα την υπεσπιστεί. Το Μάρτιο θα πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία για να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο τη περιφερειακή πολιτική επί τόπου. Σα ευχαριστώ. Much, uh... Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νοβάκοφ και ο διεισηγητή. Πρόκειται για την έκθεση ε, αντικτύπου, είναι έκθεση υλοποίηση και όχι εκτίμηση για το μέλλον. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις εφαρμογής, η Επιτροπή μας έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Γιατί πέρα από την εκτίμηση και την αξιολόγηση των όσων έχουν ήδη γίνει, μας δίνει μοναδική ευκαιρία να δώσουμε και συστάσεις και συμβουλές για το μέλλον. Νομίζω ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι μια τέτοια περίπτωση, ιδιαίτερα τώρα, κατά το Brexit. Και έχω τεράστιες ελπίδες από την έκθεση αυτή και τις ε, συνέπειες. Χαίρομαι που συνεργαζόμαστε με τον Derek Βον, ο οποίος είναι πολύ πρόθυμος να δεχτεί τις ε, όποιες προτάσεις μας. Μπορούμε πολιτικά λοιπόν να αξιοποιήσουμε την έκθεση για να πούμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά τη πολιτικής συνοχή ιδιαίτερα σε τέτοιες περιφέρειες. Σε λίγους μήνες θα συζητήσουμε το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα υπόλοιπα της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει λοιπόν πιστεύω η έκθεση να στείλει ένα μήνυμα ότι υπάρχουν περιφέρειες όπως η Βόρεια Ιρλανδία που κάνουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά για τη ζωή των ανθρώπων τέτοια ταμεία όπως είναι τα ταμεία συνοχής. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όλα αυτά. Πέρα από τα συναισθηματικά και τα πολιτικά και όλο αυτό το βάρος που νιώθουμε ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή και το ξαναλέω λόγω του Brexit αν είμαστε τελείως νυφάλιοι και αντικειμενικοί, νομίζω η πολιτική συνοχή στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ένα γνήσιο παράδειγμα. Ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Ειδικά στο δικό μας τομέα της περιφερειακής πολιτικής και δεν μπορούμε να δώσουμε υποστήριξη με χρηματοδοτικά μέσα αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας ΕΣΠΑ κάθε φορά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Για να δούμε λοιπόν την έκβαση της έκθεσης, αλλά έχω τεράστιες προσδοκίες, επαναλαμβάνω, και ελπίδες να αποθέσεις αυτή. Και ο Ντέρεκ ε, θέλει όσο γίνεται περισσότερο να το επικοινωνήσει αυτό, να, να το εκπέμψει ως μήνυμα και εκτός Επιτροπής μας για να δούμε τι, έχουν γίνει όλα, τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος σκιώδης. Ο κ. Βαν Μίλτενμπερg, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Uh, Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη εξ ονόματο του δικού μα σκιώδου σύγητου. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί πολλά σημαντικά ήδη υπόθηκαν από προλαλήσαντε. Θέλω μόνο να προσθέσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, όχι απλώς να επικεντρωθούμε στο πρόγραμμα για την ειρήνη peace, αλλά και το Interreg για να δείξουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία που έφερε η Ευρώπη στη Βόρεια Ιρλανδία και από αυτή τη σκοπιά. Και επίση θα ήθελα να κοιτάξουμε και το μέλλον βεβαίως βάσει των ε, σημερινών προγραμμάτων να δούμε πώς η διασυνορική συνεργασία θα μπορούσε και στο μέλλον να γίνει, να μάθουμε από την εμπειρία, από τα παραδείγματα του παρελθόντος και στο μέλλον μετά το Brexit. Διότι ένα είναι βέβαιο. Είτε κανείς συνεργάζεται στην Ευρώπη, εντό τη Ευρώπη, μεταξύ των περιφερειών και οπότε έχει το ίντερεκ. Αλλά όταν είσαι τρίτη χώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει η διασυνορική συνεργασία. Ε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ η κυρία Άντερσον. Ε, ευχαριστώ. Να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Τερεκβόν για την πρωτοβουλία αυτή και που μας δίνει μια ευκαιρία να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η Επιτροπή έχει επικεντρωθεί στον αντίκτυπο που είχε η πολιτική συνοχή στη Βόρεια Ιρλανδία. Είναι ένας, μια περιοχή που γνωρίζω πολύ καλά, προέρχομαι από μια πόλη που λέγεται Ντάρι και υπάρχουν πάρα πολλές ε, οργανώσεις ε, ε, και έχουμε και τον ε, τομέα τον κοινοτικό, πολλές μικρές και μεσές επιχειρήσεις, ε, υποδομές που αναπτύχθηκαν, άνθρωποι που έχουν επωφεληθεί και είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την συνεισφορά της Ευρώπης στην οικοδόμηση της ερευνητικής διαδικασίας με έναν τρόπο που κανένα άλλο πρόγραμμα και κανένα άλλο ταμείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε τέτοιο αντίκτυπο. Το 10% του ΑΕΠ της Βορειας προέρχεται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, είμαστε καθαροί δικαιούχοι. χωρίς ε, αυτό το προϋπολογισμό δεν θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει ούτε η κυβέρνηση και είχε πάρα πολλέ ε, ευκαιρίε να χρησιμοποιήσει την συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλά προγράμματα και υποδομές θα μπορούσε να αναφερθεί κανεί, αλλά προέρχομαι από τον Τέρι και παίρνουμε το χάρη εκεί υπάρχει μια γέφυρα της ειρήνης η οποία ε, ουσιαστικά οικοδομήθηκε ως ε, συνέπεια της χρηματοδότησης ε, για την ειρήνη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ουσιαστικά υπήρχε μια μειοψηφία το 20% του πληθυσμού ήταν, είχε τον έλεγχο της πόλης, ήταν στο Συμβουλίο ενώ όσοι προερχόμασταν από την κοινότητα ουσιαστικά ε, έπρεπε να να μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση για να έχουμε ένα σπίτι και όταν ε, τελικά χτίστηκε αυτή η γέφυρα της ειρήνης ήταν μια από τις ε, πρωτοβουλίες που βοήθησε την ένωση της πόλης. Υπήρχε μια διαιρεσμένη πόλη από το νερό Είχαμε την άλλη πλευρά της πόλης ε, με την ε, κοινότητα των ενωτικών και υπήρχε μία σύνδεση και τότε σκέφτηκαν ε, οι άνθρωποι ότι αυτή η γέφυρα Πώ ήταν άχρηστη, δεν μπορούσε να περάσει αυτοκίνητο από εκεί. Ποιο ήταν ο σκοπό, όμω ήταν ένα σύμβολο, μια συνδεση και τοτε σκεφτηκαν οι ανθρωποι οτι αυτη η γεφυρα όπως ηταν αχρηστη δεν μπορουσε να περασει αυτοκινητο απο εκει Ποιος ηταν ο σκοπο όμως ηταν ενα συμβολο μια εικονα των υποδομών της ειρηνευτικής διαδικασίας που έκανε πολύ μεγάλη διαφορά στην συνένωση των κοινοτήτων. Έτσι λοιπόν ε, θα ε, ε, έλεγα ότι είχαμε διάφορες μικρές ομάδες, μικρές και μεσές επιχειρήσεις που ε, ουσιαστικά υποφελήθηκαν από τη χρηματοδότηση και έγινε τρομερή δουλειά σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι άνθρωποι βλέπουν τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία. Ε, μέσα από τα διάφορα προγράμματα, το PIS 1, 2, 3 και τώρα μέσα από το PIS 4. Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά ε, καθώς βλέπουμε τον αντίκτυπο και εξετάζουμε τα ζητήματα που έθεσε ο εισηγητής, ε, όλα αυτά θα παρουσιάσουν στους ανθρώπους γιατί ένας από τους λόγους που υπάρχει πραγματική ανησυχία και εδώ διαφωνώ με τον κύριο Φλακ είναι ότι με κάποιο τρόπο θα διαιρέσεις ε, ε, αυτό που έχουμε πετύχει στο Βορρά και υπάρχει φυσικά φόβος από τους ανθρώπους ε, που θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής ε, και ε, λόγω της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πολιτικής συνοχής. Δεν φαντάζομαι ότι ο κύριος Βον θα μπορέσει να διαχωρίσει τον Brexit και τις επιπτώσεις του Brexit στη Βόρεια Ιρλανδία από την έκθεση αυτή. Θα ήταν καθαρή τρέλα να προσπαθήσουμε να το γνωρίσουμε αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν θεσπίσει προγράμματα και φυσικά προγράμματα που ισχύουν πολύ πέρα από το 2020 και δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχουμε περάσει μια μεταβατική περίοδο και έληξε η εποχή της σύγκρουσης και περάσαμε σε μια κοινωνία που το έχει αφήσει αυτό πίσω. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα και η πολιτική συνοχή στη χρηματοδότηση για την ειρήνη έχει συνεισφέρει τα μάλα σε αυτό. Μόλις πριν λίγους μήνες είχαμε ειδικά ε, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, ήρθαν άνθρωποι εδώ στις Βρυξέλλες που μας παρουσίασαν κάποιες μικρές περιπτώσεις και μπόρεσαν να δείξουν στους βουλευτές και σε άλλους την σημασία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση της ερνευτικής διαδικασίας. Είτε πρόκειτο ε, για ένα νοσοκομείο στην πόλη μου όπου ε, δημιουργήθηκε μια μονάδα ε, ραδιοθεραπείας, είχαμε ομάδες προεμφυλακισμένων και τελικά μπορέσαμε ουσιαστικά να ενώσουμε ε, τους ανθρώπους ε, στον τεριμέσο αυτού του νοσοκομείου. Δεν θα είχαμε μονάδα ραδιοθεραπείας στο νοσοκομείο Γκάβιν αν δεν είχαμε τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την υποδομή που χρειαζόταν ε, πάρα πολύ Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από ε, πρώην ε, που ε, κάθονται και συζητούν, άνθρωποι που κάθονται στην, ε, ίδια, στο ίδιο δωμάτιο και συζητούν, κάνουν δύσκολες συζητήσεις. όλα αυτά συνέβησαν λόγω της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην αφήσετε σε κανένα να πει σε αυτή την Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε ρόλο να διαδραματίσει στην πολιτική διαδικασία, στην ειδευτική διαδικασία και στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ε, υπάρχουν τεράστιος όγκος αποδείξεων στην ε, Βόρεια Ιρλανδία που δείχνει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι λοιπόν που θα λάβει χώρα η αποστολή και νομίζω ότι θα τα δείτε κι εσείς με τα μάτια σας, θα συζητήσετε με ανθρώπους εκεί επί τόπου και χάρηκα από ξετροσυγητή τον και άλλους να λένε ότι ε, χάρη ε, πρέπει να πούμε ότι έχει εμπλακεί η κοινότητα στην ε, εφαρμογή των διαφορών προγραμμάτων ήταν καθοδηγούμενα από την κοινότητα. Ελπίζω λοιπόν όταν θα πάμε στο Βορρά, στη διερευνηστική αποστολή, ε, θα δοθεί στους ανθρώπους ευκαιρία να εξετάσουν ε, την εφαρμογή της χρηματοδότησης, ε, του ίντερεγ, της πολιτικής συνοχής στη Βόρεια Ιρλανδία και στην ίσο της Ιρλανδίας. Οι άνθρωποι θα δουν με τα ίδια τους τα μάτια και ουσιαστικά ε, η περίπτωση του να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διευθέτηση για να ε, μείνει η Βόρεια Ιρλανδία ε, στην θα δουν οι άνθρωποι ε, πόση ζημιά μπορεί να γίνει αν αφαιρεθεί ε, αυτή η χρηματοδότηση συνοχής γιατί η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στο να υπάρχει ανάπτυξη σε όλη την Ιρλανδία ε, μέσω του ίδιου τρόπου όπως χρηματοδοτεί η πολιτική συνοχής εξακολουθούμε να έχουμε ένα μακρύ ταξίδι, ένα μακρύ δρόμο, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει το ρόλο της. Έχουμε κάνει ένα δύσκολο ταξίδι και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις επιπτώσεις του Brexit στη ζωή των ανθρώπων ως συνέπεια ε, της ε, απόσυρσης όχι απλώς μιας οικονομικής στήριξης αλλά το τι σημαίνει η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους ανθρώπους που είχαν μια εμπειρία συγκεκριμένη με την κυβέρνηση. Αυτό διαφέρει πάρα πολύ από αυτά που μπορεί να προσπαθήσουν άλλοι να αποδείξουν που κατά πολλούς τρόπους δεν είναι ευχαριστημένοι. Πολλοί άνθρωποι έχουν πραγματικούς φόβους και πιστεύουν ότι αν λείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ε, δεν υπάρχει ο σημείο αναφοράς, το οποίο μπορούν να απευθυνθούν και ο πληθυσμός 1,8 εκατομμύρια αν ε, το αφαιρέσει το δικαίωμα ε, να έχει ε, Ιρλανδικό διαβατήριο γιατί 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να έχουν αυτό και αυτό σημαίνει ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι ζωτική σε αυτή τη χρονική συγκυρία και σας ευχαριστούμε κύριε Βόν που παίρνετε αυτή την ε, πρωτοβουλία και έρχεται φως ε, σε έναν ε, τομέα που θα αποκαλύψει σε αυτήν την Επιτροπή την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στην Ιρλανδία και κυρίως στο Βορρά λόγω της στήριξης που δόθηκε μέσω της χρηματοδότησης συνοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριο Ρέινκε, ο επόμενο κοιόδης. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ρέινκε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κατάγομαι από μια περιοχή η οποία έχει ε, προκλήσει προκλήσεις ε, σε μια βιομηχανή περιοχή και παρόλο που, βρίσκομαι, που βρίσκεται σε μια σχετικά πλούσια χώρα όπω είναι η Γερμανία, ε, όταν ε, μιλάω με τους ανθρώπους σε περιφερειακό επίπεδο όλοι μα λένε πόσο σημαντικό είναι να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο σε διασυνοριακό επίπεδο αλλά και σε σημεία τα οποία αναφέρθηκαν υπάρχουν ορισμένα ε, προγράμματα ε, τα, όπου τα ε, ευρωπαϊκά χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα από ό,τι τα χρήματα από το κράτος τα οποία δεν θα υπαρκούσαν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πιστεύω ότι η περιοχή καταγωγής μου συγκρίνεται με την Ιρλανδία. Μιλώντας με πολίτες εκεί πέρα οι άνθρωποι λένε ότι χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωση πολλά προγράμματα δεν θα ήταν εφικτά. Και γι' αυτό το λόγο ε, θα ήθελα να πω ότι αυτή την ε, περίοδο τα ε, χρήματα των διορθωτικών ταμπίων, τα οποία έχουν επενδυθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βοηθήσει 6.000 επιχειρήσεις ενέρχονται στα 300 εκατομμύρια ευρώ θα δημιουργηθούν ε, ε, πολλές εργασίας έχουμε 210 εκατομμύρια, 210 εκατομμύρια ε, ε, ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία θα βοηθήσουν τις κοινωνικές ανισότητες. Αναφερθήκαμε επίσης στο πρόγραμμα PIS ε, ε, για αυτήν ε, την περίοδο. Έχουμε 270 εκατομμύρια τα οποία θα επενδυθούν σε διάφορα προγράμματα συμφιλίωσης και τα τελευταία χρόνια δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε αυτόν τον τομέα και έχει αναφερθεί το πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό. Εξετάζοντας λοιπόν την επιρροή των ε, των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρο. Κάποιοι συναδέλφοι ανέφεραν ότι θα είναι δύσκολο από εμά ε, να πάμε σε, να κάνουμε μία αποστολή ε, για να μάθουμε από τους πολίτες τι κέρδισαν στο παρελθόν και τα προβλήματα και τις ανησυχίες που μπορεί να έχουν για το μέλλον με αφορμή το Brexit. Για μένα είναι δύσκολο λοιπόν το πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό και γι' αυτό θεωρώ ότι επίσης θα πρέπει να έχουμε αότα σχετικά με τι ανησυχίε που υπάρχουν εκεί πέρα καθώ καθώς επίσης και με το ρόλο τον οποίο θα πρέπει να παίξουμε εμείς, ούτως ώστε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια να μην ε, χαθεί. Υποστηρίζω απόλυτα λοιπόν το σημείο ότι ναι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην επιρροή, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εξετάσουμε και το μέλλον και ως ε, ειδική στην περιφερειακή ε, χρηματοδότηση στην Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις κοινότητες της Βόρειας Ιρλανδίας ε, και στο μέλλον ό,τι και αν συμβεί με, όπως και αν είναι το ε, Brexit. Ε, έχουμε λοιπόν να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το σημείο. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό το ε, θέμα. ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νταμάτο. Ευχαριστώ. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για ιστορικές περιοχές, κοινωνικές, πολιτικές και φυσικά θίγονται από τις διαπραγματεύσεις ε, το Brexit. Ε, είχαμε το PIS 3 την περίοδο 2007-2013, ε, το οποίο ενίσχυσε την πρόοδο προς μια σταθερή και ειρηνευτική κοινωνία και ήθελε να προωθήσει τη συμφιλίωση μεταξύ της Βορειάς Ιρλανδίας και των όμορων περιοχών. Το πρόγραμμα είχε στόχο την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και διαθέτει μια προοικοδότηση 330 εκατομμύρια ευρώ. Τα 220 προέρχονται από το ΕΤΠΑ Φαντάζομαι ότι η τελική έκθεση ε, του 2017 ε, θα πρέπει να συμφτεί. Έτσι λοιπόν θέλουμε να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα του προγράμματος και νομίζουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο σχέδιο της έκθεσης. Στο σημερινό προγραμματισμό υπάρχει ένα άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Βόρεια Ιρλανδία και ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα Interreg ε, για άδαφη και συνεργασία μεταξύ της Δημοκρατίας Ιρλανδίας, Βρετανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, εμείς ε, θέλουμε και τα δύο προγράμματα να υλοποιηθούν ως το τέλος. Οι διαπραγματεύσεις για τον Brexit είναι πολύ δύσκολες, όμως ε, Κυρίω ε, ω Ευρωπαίοι πολίτη, θέλω να πω ότι όποιο και αν είναι το τελικό αποτελέσμα των διαπραγματεύσεων, δεν θα πρέπει να επιστρέψουμε στη βία που χαρακτήρισε τα 30 χρόνια από τα τέλη τη δεκαετία του 60 στο τέλη τη δεκαετία του 93.000 3.000 ε, θάνατοι, ε, σοβαρή θρησκευτική και πολιτική σύραξη στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να τα επιτρέψουμε. Ε, και χάθηκε και η Ντολόρες ε, Γιορτάν ε, η οποία ήταν καταπληκτική τραγουδίστρια και είχε τραγουδήσει το τραγούδι «Ζόμπι» και αφορούσε τη βία που επιδεικνύουν οι άνθρωποι. Τα ζόμπι είναι οι ζωντανοί νεκροί, αυτοί που δεν βλέπουν και έχουν συνηθίσει στη βία. Η πολιτική συνοχής ουσιαστικά μας βοήθησε και να ε, κλείσουν κάποιες πληγές. Brexit είτε όχι, όλα θα πρέπει να γίνει για να μην επαναληφθούν πλήρως ε, αυτές οι σκηνές ε, των παιδιών που πεθαίνουν λόγω μια έκρηξης βόμβας, η εικόνες των τάξη που κυκλοφορούν στους δρόμους. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα όνομα στη λίστα που θα ήθελε να μιλήσει ο κύριος ε, Ράπε. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα στα πλαίσια της Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και γενικότερα στην πολιτική συνοχής. Προσωπικά νομίζω ότι η Βόρεια Ιρλανδία είχε την ευκαιρία να επωφεληθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής και τα αξιοποίησε θαυμάσια με πολύ καλή διαχείριση, με συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό σήμερα και ξεκάθαρα και να εξηγήσουμε σε κάποιους άλλους για ποιο λόγο ε, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική συνοχή για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι χρησιμεύει. Εγώ έχω διατελέσει δήμαρχος. Και στη συνέχεια περιφερειάρχης, σε μια περιφέρεια στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ξέρω τι θα πει λοιπόν να είσαι περιφερειάρχης σε μια παραμεθόρια περιοχή και ε, όλες αυτές οι περιφέρειες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους και τη σημασία τους και χρειάζονται βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές είναι κρίσιμη και κομβική. Έχουμε λοιπόν μια σχετική πείρα. Ε, τώρα αυτό θα πρέπει να κάνουμε ε, να σκεφτούμε το μέλλον. Τι θα γίνει. Η σημερινή πολιτική συνοχή έτσι όπως ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήσιμη συμπεριλαμβάνει αρκετά ε, τους ενδιαφερόμενους τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί σε κάποιες χώρες η πολιτική αυτή είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτική. Άρα, τι πολιτική συνοχή είναι αυτή που χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να μας προβληματίζει και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχει περισσότερο ο πληθυσμός, ή τοπικές κοινωνίες για να γνωρίζουν πραγματικά ότι ε, αξιοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια, χρήματα των ε, φορολογουμένων για να λύσουν δικά τους ζητήματα. Καμιά φορά η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει την ίδια οπτική γωνία. Το πρόγραμμα Leader ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και στο μέλλον θα πρέπει ενδεχομένως να προβλέψουμε ένα σχετικό πρόγραμμα Leader για τους Δήμους και τις κοινότητες δηλαδή να καταβάλλονται τα χρήματα σε έργα όπου συμμετέχει η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικές επιχειρήσεις για να μπορεί ο κόσμος να λύνει τα τοπικά προβλήματα σε τοπικό επίπεδο και όχι σε κεντρικό. Αυτά μπορεί να φαίνονται ε, λεπτομέρειες από μακριά αλλά όταν είσαι επιτόπου μπορεί να είναι ένα τεράστιο ζήτημα για τους ντόπιου έτσι θα συμμετέχει περισσότερο ο κόσμος, η τοπική κοινωνία επαναλαμβάνω και θα ε, καταλαβαίνει, θα καταλαβαίνει καλύτερα και θα κάνει κτήμα του ε, την πολιτική αυτή γιατί αφορά τα καθημερινά του προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Γκονζάλες ε, Χερνάντες ε, από τη Γενική Διεύθυνση Γυρίγιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα. Η Κομισιόν θα ήθελε να ευχαριστήσει την Επιτροπή ε, για, το, για την ενδιαφέρουσα αυτή συνεισφορά σχετικά με τη Βόρεια Ιρλανδία. Υπήρξαν πάρα πολλέ σημαντικέ συνεισφορέ και έχει γίνει πολύ σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διάφορα προγράμματα, τα κοινωνικά ταμεία, αγροτικά κοινοτική χρηματοδότηση μιλάμε για 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ μονάχα από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, ε, και έχουν υπάρξει και από άλλα ταμεία σημαντικές ε, συνεισφορές πέρα από τα προγράμματα Peace και Interact επίσης θα θέλαμε να αναφερθούμε ε, στη χρηματοδότηση που γίνεται στην υποστήριξη επιχειρήσεων όπου η Βόρεια Ιρλανδία είναι πάρα πολύ καλή σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς επίσης και σε τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα η Επιτροπή λοιπόν έχει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει επίσης διασυνοριακά προγράμματα ε, τα οποία ε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αλλαγή στην περιοχή. Ε, επίσης, επενδύουμε στην υγεία όπως αναφέρθηκε από την κυρία Άντερσον και ε, σε άλλου ε, τομεί που διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων στην περιοχή και τέλο, φυσικά τα προγράμματα PIS ε, τα οποία γνωρίζουν τα μέλη τη Επιτροπή, γνωρίζουν την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το PIS ένα πρόγραμμα όπω κανένα άλλο εργαζόμαστε σε μια περιοχή διαμάχη. προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τι κοινωνίε που αντιμάχονταν για πάρα πολύ καιρό και θέλουμε, δεν θέλουμε να στομπιεύσουμε μονάχα ανθρώπου οι οποίοι συμμετείχαν στη διαμάχη και σε νέους ανθρώπους ε, μέσω της εκπαίδευσης ε, κοινών χώρων, ε, θέματα τα οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν και μελλοντικά τη Βόρεια Ιρλανδία και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Βόν και άλλα μέλη για να μπορέσουμε να παράσχουμε την υποστήριξη την οποία χρειάζονται για το συγκεκριμένο σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Βόν τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τις συναδέλφους ε, για τις συνεισφορές τους ε, και ε, θα ξεκινήσω απαντώντας για το ζήτημα του Brexit αφορά την εφαρμογή. Αν δεν λέγαμε ότι το, το θέμα είναι η εφαρμογή, τότε δεν θα είχαμε την άδεια να κάνουμε αυτό το σχέδιο. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι καθώς ε, θα ε, συντάσουμε την έκθεση, καθώς θα κάνουμε τις επισκέψεις, θα εξετάσουμε το όφελος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τη Βόρεια Ιρλανδία και θα δούμε και παραδείγματα πάνω σε αυτό εάν ε, δεν είχαμε την εργασία πάνω σε αυτό ε, θα μπορέσουμε να εργαστούμε, θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε πάνω σε αυτό. Επίσης, ε, θα δεν θα πρέπει να ε, έχουμε γρήγορα συμπεράσματα, θα πρέπει να εξετάσουμε τα παραδείγματα, να δούμε ότι είναι σημαντικό να το τι θα γίνει σε περίπτωση που αποχωρήσει το, η Μεγάλη Βρετανία Ε, θα μιλήσουμε για τις ε, συνέπειες ε, του Brexit πάνω σε αυτή την έκθεση, στο πλαίσιο όμως το οποίο μόλις έθεσα. Επίσης αναφέρθηκε η σημασία να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό ενώ και η Κομισιόν το ανέφερε αυτό Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν όλα αυτά, να δούμε τις ε, συνεργίες οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των διαφορών προγραμμάτων PIS, ε, Interact ε, και των υπολείπων για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το μέλλον. Η Μαρτίνα ανέφερε την σημασία να εξετάσουμε πρακτικά παραδείγματα μεταξύ των έργων των οποίων αναφέρθηκαν προηγουμένως και επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε πρακτικά παραδείγματα ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τα μικρότερα σχέδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μερικές φορές επικεντρωνόμαστε στα ε, μεγάλα ποσά, στην αύξηση του ΟΕΠ, στα μεγάλα σχέδια. Όμως πολύ συχνά η διαφορά στις κοινότητες και στους ανθρώπους είναι τα μικρότερα σχέδια. Έχουμε δει κάποια τέτοια παραδείγματα και θα πρέπει να επικεντρωθούμε πάρα πολύ, ε, να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο πάνω σε αυτά τα μικρότερα σχέδια, να συζητήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα τα προγράμματα, να δούμε ποιοι έχουν υποφεληθεί από όλα αυτά και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην έκθεσή μας ε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας ε, και επίσης ε, θα έχουμε μαθήματα από όλο αυτό ε, σχετικά με το πώς θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε την πολιτική μας για μετά το 2020 διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι κοινότητες και τα μεμονωμένα άτομα παίζουν ένα ρόλο στην ανάπτυξη και στην απόδοση των περιφερειακών προγραμμάτων. Είναι ένα μεγάλο σχέδιο είναι ένα μεγάλο, το μεγάλο θέμα της ημέρας σχετικά με τον Brexit και την επιρροή που θα έχει στη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όμως αυτό και να μας βοηθήσει ούτω ώστε να βελτιώσουμε την περιφερειακή μας πολιτική για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο, ε, τα επόμενα βήματα για την έκθεση θα είναι η ε, οργάνωση επιτροπής για την ε, Μεγάλη Βρετανία, για, 20, για τη Βόρεια Ιρλανδία, για 21-22 Φεβρουαρίου εγκρίθηκε Μαρτίου ε, θα εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων και μπορούμε να, ξεκινήσουμε το έργο μας πάνω σε αυτό και στη συνέχεια η, η ε, έκθεση θα προετοιμαστεί λαμβάνοντας υπόψη ε, τις απόψεις ε, που θα έχουν ακουστεί εδώ πέρα καθώς επίσης και από την αποστολή που θα γίνει ενώ τους επόμενους μήνες μετά τις διακοπές του καλοκαιριού θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα θέσει ο κ. Βαν πριν Ο κ. Φλακ χωρίς μικρόφωνο. Just on a clear point. Ε, για να διευκρινίσω κάτι. Ο κύριος Βον, συνοψίζοντας, είπε αν αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα μην έχετε καμία αμφιβολία. Θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο 29 Μαρτίου 2019. Θα συμβεί. Μην αμφιβάλλετε και μην σας μπαίνουν τώρα αμφιβολίες. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκρίνηση. Εγώ παραμένω στο εάν, πρόεδρε, λέει ο κύριος Βον. Καλά, ο καθένας έχει την προσωπική του και την πολιτική του θέση. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να έχουμε μια πάρα πολύ καλή έκθεση ε, για την εφαρμογή και τον αντίκτυπο. Ωραία. Κλείνει η συζήτηση για αυτό το θέμα εδώ ενδιαφέρον θα έχει να δούμε την έκθεση στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, προχωρούμε στο επόμενο θέμα, στη μέση διάταξη, που είναι... This is uh, the uh, opinion. Είναι γνωμοδότηση ε, με συντάκτη τον κύριο Ντάνιελ Μπούντα. Ε, είναι η έκθεση για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι επί της ουσίας αρμόδια και κάνει την έκθεση. Εμεί κάνουμε γνωμοδότηση ε, νομοθετικού περιεχομένου. Το λόγο έχει πρώτο συντάξει νομοδότησης και μετά οι υπόλοιποι σκιώδε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόταση τροποποίησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα την προσπάθεια του Επιτρόπου Στυλιανίδης Στυλιανίδη να υιοθετήσει την πρόταση αυτή. Η πρόταση αυτή καθόρισε μια συνάντηση που έγινε στις 16-17 Ιανουαρίου των Γενικών Διευθυντών Πολιτικής Προστασίας 10 κρατών μελών Γερμανία, Κροατία, Κύπρος, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία Πορτογαλία, Τσεχία και Ρουμανία. Εκεί ε, χαιρέτησαν αυτή την πρόταση δηλώνοντας την δυνατότητα να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων. Ε, η γενικοί διευθυντέ ε, ασχολούνται με το θέμα τη αντιμετώπιση των καταστροφών. Αυτό ο μηχανισμό πολιτική προστασία αποτελεί στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντά ταχύτατα σε περιπτώσει έκτακτη ανάγκη που μπορεί να λάβουν χώρα και εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτρέψουν ε, μια συντονισμένη παροχή βοήθεια ε, μέσω τη συγκέντρωση των πόρων από όλα τα συμμετέχοντα μέρη, ανθρωπιστικέ κρίσει, τις ε, πυρκαγιές, ε, τυφώνες, καταιγίδε, αλλά και πλημμύρες ε, και οι σεισμοί των τελευταίων ετών έχουν επιβάλει αλλαγές στην νομοθεσία σε σχέση με την πολιτική προστασία επιπρόσθετα έκτακτες καταστάσεις που έχουν πλήξει πολλά κράτη-μέλη έτσι ώστε να οδηγούν στο να είναι εντελώ απαραίτητο να δίνεται αυτή η αμοιβαία βοήθεια ε, στην περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους την ε, κρίση και χρειάζονται μια συντονισμένη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν προτείνει μια σειρά νέων στοιχείων που έχουν ε, ως αντικείμενο την παγίωση των ικανοτήτων της πρόληψης αλλά και του συσχετισμού με καλύτερο τρόπο με τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει με την ενδυνάμωση των συλλογικών τεχνικών ικανοτήτων ε, για να απαντηθούν οι περιπτώσεις ε, κρίσης. Το Rescue θα έχει ένα υποστηρικτικό ρόλο στην περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση και θα διασφαλίσει συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών. Και θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση στις συζητήσεις που είχαν αυτοί που ασχολούνται με την διαχείριση των καταστροφών. Υπήρχε ε, μία ερώτηση ποιος θα συντονίσει αυτή τη δομή, αν ε, ε, είναι ο συντονισμός από την Κομισιόν ή αν θα εμπλακούν και τα κράτη-μέλη. Η δική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται στενή συνεργασία σε αυτό το τομέα. Και επίσης από την πλευρά των διευθυντών υπήρχε μια παρατήρηση σε σχέση με την ε, ανάγκη ο κατάλογος των μέσων που προτείνεται να είναι κάτι ευέλικτο και όχι να είναι περιοριστικός ο κατάλογος γιατί μπορεί να παρουσιαστούν συγκεκριμένες ε, ανάγκες. Θεωρώ ότι οι προτάσεις της Κομισιόν είναι πολύ σημαντικές και απαντούν πλήρως ε, στις πρόσφατες προκλήσεις. Στο έγγραφο εργασίας θα επικεντρωθώ σε κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, που ε, ουσιαστικά σχετίζονται με τη συνεισφορά των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και στην πρόληψη των κινδύνων και στη διαχείριση των κρίσεων. Είναι απολύτως απαραίτητη η αύξηση των συνεργειών μεταξύ των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων ιδίω η συμπληρωματικότητα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Οι εξάντε προϋποθέσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ε, ότι οι επενδύσεις μέσω των διαφορετικών ταμείων θα ανταποκρίνονται ε, στα αιτήματα για την αντιμετώπιση κινδύνους. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στην ε, πρόληψη των καταστροφών όπως σημαντική είναι και η ε, παγίωση αντίδραση στην περίπτωση κρίσης, γιατί η τοπική αυτοδίκηση είναι η πρώτη που μπορεί να παρέμβει σε τέτοιες καταστάσεις. Η ειδική προετοιμασία και η καινοτομία είναι ουσιαστικές επιτυχές της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να έχουμε πιο αποτελεσματικές δράσεις και για να παγιωθεί ο διάλογος μεταξύ των κρατών μελών. Εδώ βλέπω σημαντικό ρόλο των κέντρων αριστείας και των πανεπιστημίων που μπορούν να κάνουν έρευνα σε μηχανισμούς προστασίας που παρεμβαίνουν ταχύτατα. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο πρόληψης κατά των καταστροφών μέσω της προετοιμασίας του αρμόδιου προσωπικού και μέσω του συντονισμού τους ε, στην ε, περίπτωση των ειδικών εφεδρικών μονάδων. Ε, το θέμα της γνώσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και δράσεις προετοιμασίας εθελοντών οι οποίοι δρούν σε απομονωμένες περιοχές ε, και περιορισμένης πρόσβασης ακριβώς ε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Στη Ρουμανία, παραδείγματος χάρη, είχαμε ένα αεροπορικό ατύχημα και οι πρώτοι που παρενέβησαν ήταν οι πολίτες ε, και όχι οι αρχές γιατί οι πολίτες ήξεραν ακριβώς τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Και τέλος κάποιες τεχνικέ λεπτομέρειες. Ε, η έκθεση, όπως είπατε και εσείς, ε, Πρόεδρε, ε, ουσιαστικά θα είναι αρμόδια η Επιτροπή ΕΝΒΗ για την έκθεση αυτή. Εμείς θα έχουμε κάποιες τροπολογίες που θα προτεθούν και φυσικά περιμένω και τη συνεισφορά όλων των συναδέλφων αλλά και κυρίως των σκιωδών εισηγητών για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Thank you very much. Now I'll give the floor to the... Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο σκιώδης Η ε, κυρία Ροντρίγκες πρώτη. Ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζουμε τις τεράστιες ε, φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές καταστροφές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν ε, χαθεί ε, πολλές ζωές και έχουμε καταστροφικές επιχειρήσεις για τις επιχειρήσεις, για το περιβάλλον και για την πολιτιστική κληρονομιά. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνο του. Αυτές οι καταστροφές, οι πυρκαγιές του 2017 ήταν σύμπτωμα όμως ε, το σύστημα απάντησης ε, επίσης ε, μας έδειξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν καθυστερήσεις. Βλέπουμε σημαντικές ελλείψεις ως προς τους διαθέσιμους πόρους οι εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών δεν ήταν επαρκείς. Επομένως, χρειαζόμαστε έναν ένα δεσμευτικό κανονισμό που να ε, μας διευκολύνει να απαντήσουμε σε ορισμένα είδη καταστροφών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την κατάλληλη στιγμή. Θα πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο σύνολο υποχρεώσεων των κρατών μελών σε περίπτωση ε, φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και η συνθήκη της Λισαβόνας μας επιτρέπει να προχωρήσουμε ε, μέσω της ρήτρα αλληλεγγύης. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να σεβαστούν τις υποχρεώσεις παροχής αλληλεγγύης ε, καλύπτοντας τα υφιστάμενα κενά κυρίως σε ό,τι αφορά στον εθελοντικό χαρακτήρα παροχής της βοήθειας. Η Επιτροπή μας έχει σημαντικό ρόλο στην έκθεση αυτή προκειμένου να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις και πραγματική διάρθρωση με τις ε, σχετικές πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με μέτρα πρόληψης των καταστροφών και ε, καλύπτοντα θέματα υγείας και μετανάστευσης, αλλά και φυσικά και καλύπτοντα και θέματα έρευνα και κοινοτομίας. Ε, η περίπτωση ε, της ε, σοσιαλιστικής ομάδας ε, θέλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πρόληψη και κατάρτιση των ομάδων. Στην περίπτωση της κατάρτισης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και ε, θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των διευθυντών για τις διάφορες καταστροφές. Επίσης, ε, θα πρέπει να έχουμε δουλειά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός και διάρθρωση με τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά την απάντηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και Επίσης, ενίσχυση αυτού του μηχανισμού σημαίνει να αναγνωρίσουμε τη σημασία των κρατών ε, μελών, αλλά και τις ε, δυσκολίες, ε, αλλά και να ανταποκριθούμε στο αίτημα της αλληλεγγύης αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια συμφωνία ε, μεταξύ μας για να προστατευτούν οι Ευρωπαίοι αλλά και μη Ευρωπαίοι πολίτες. Ε, χρειάζεται ένα αποθεματικό, μια εφεδρική μονάδα πολιτικής προστασίας. Αυτό το δίκτυο βέβαια δεν θα αντικαταστήσει τις ε, εθνικές μονάδες αλλά θα αποτελεί μια αποτελεσματική μονάδα απάντησης στις πιο δύσκολες συνθήκες και στις πιο δύσκολες καταστροφές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει σκιώδηση Τρεις από το ΙΣΙΑ, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, όχι. Ο κύριος Γιάκοφσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω μερικά πράγματα από πλευρά μου. Δυστυχώς έχω και εγώ εμπειρίες με ορισμένες δυσάρεστες καταστάσεις θεομηνίες, φυσικές καταστροφές όπως είναι δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες. Είναι πολύ σημαντική και πάρα πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και βέβαια θα αγωνιστώ πάρα πολύ να υπάρξει καλό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει να φροντίσουμε, να κοιτάξουμε στο μέλλον πώς θα δρούμε ταχύτερα και αποτελεσματικότερα και πώς θα αντιδρούμε σε τέτοιες έκτακτες ε, καταστάσεις κατεπίγουσες που αντιμετωπίζουν οι γειτονικέ μας χώρες. Εκεί θέλω έναν ευρύ, ευρύτερο ε, περιφερειακό μηχανισμό. Έχουμε ήδη μακροπεριφέρειες, προσωπικά είμαι αρμόδιος για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιωνίου και θα ήθελα να δημιουργηθεί ένα κέντρο αντιμετώπισης θεομηνιών. Ξέρετε ότι στα Βαλκάνια στην Ιταλία γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Και στην περιοχή της Αδριατικής μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κέντρο και η μακροπεριφέρεια να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση και της συγκεκριμένη πολιτικής. Διότι είναι πολύ πιο απλό να πάει κανείς από την Ιταλία ένα αεροπλάνο πούμε, να έρθει στη Δαλματία ή στην Πούλα να σβήσει να σβήσει μια φωτιά ή να βοηθήσει σε περίπτωση σεισμού πλημμύρας. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση αυτό, ε, αλλά πρόκειται πάλι για χρήματα. Δηλαδή, ο μηχανισμός ε, για την χώριση κονδυλίων ε, στις πληγήσεις περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Ξέρουμε ότι σε περίπτωση φυσικής καταστροφής τα 300 ή τα 500 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό ε, που χρειάζεται συνολικά, αλλά δεν θέλουμε να το καταβάλουμε την ίδια στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιγόντως μια προκαταβολή 5 εκατομμυρίων μέχρι να αποφασιστεί τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Όταν υπάρχει μια θεομηνία, κάποια στιγμή πρέπει επιγόντως να σταλούν ε, βοήθειες και χρήματα. Είναι παράλογα αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι υπήρξε μια φυσική καταστροφή, ας πούμε, που έχει προκαλέσει ζημίες ε, της τάξης εκατομμυρίων, έχουν, έχει γκρεμίσει σπίτια ένα σεισμό στην Ιταλία και μετά περιμένουμε μήνες για να εγκρίνει τα κονδύλια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να ε, μπορεί να αντιδρά ταχύτερα. Γιατί απογοητεύεται ο κόσμο και θεωρεί ότι η Ευρώπη αδιαφορεί για το τι του συμβαίνει. Αυτές είναι οι δύο προτάσεις μου. Και ευχαριστώ και ελπίζω κάπως να βρω τη θέση τους και στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Μαγζέ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ροπέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, θέλω να συγχαρώ ε, τον εισηγητή για την ε, ε, προστασία και χαίρομαι για την πρωτοβουλία αυτή Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Η δική μα Επιτροπή έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει εδώ, γιατί σε τελική ανάλυση οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι εκείνες που φέρουν αυτό το βάρος και κουβαλάνε αυτό το σταυρό ε, υλοποίησης αυτής της πολιτικής που πολλέ φορέ μπορεί να φόρει τους. Δεν έχω πάρα πολλά σχόλια να κάνω. Είναι συγκεκριμένοι οι στόχοι της ε, γνωμοδότησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να απαριθμούμε ε, τα εργαλεία που έχουμε ή το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Γιατί έχει επιλεγεί ένα ακρονίμιο που είναι δύσκολο να προφέρουν οι μη αγγλόφωνοι θα πρέπει να προωθήσουμε την εθελοντική συνεργασία και να βοηθήσουμε το κέντρο συντονισμού. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε γραφειοκρατικές δομές ε, γενικά. Και χαίρομαι για την πρόταση τροποποίηση του άρθρου 12. Όπως έδειξαν οι δασικές πυρκαγιές πρόσφατα, χρειαζόμαστε πηγόντως ε, ε, κάποιο εξοπλισμό πυρόσβεσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρά για άλλη μια φορά στο πρόβλημα, ε, αλλά δεν αναλύει ε, τους ενδεχομένους κινδύνους και τις απειλές. Αν είχε γίνει μια τέτοια ανάλυση, ε, τότε στην νομοθετική πρόταση θα είχαμε βάλει κάποιες ρυθμίσεις για την άρση των επιπτώσεων ε, πυρηνικών ατυχημάτων. Ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες απαρχαιωμένους παλαιάς τεχνολογίας ε, που θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν και δεν θα πρέπει να αναβάλουμε την πρόληψη ε, κάποιου πυρηνικού ενδεχομένου ατυχήματος. Υπάρχουν και ανθρωπογενείς καταστροφές, δεν είναι όλες φυσικές θα πρέπει το άρθρο 12 να συμπληρωθεί με κάποιες διατάξεις σχετικά με την συνεργασία για την αντιμετώπιση και τέτοιων ε, καταστάσεων. Ας πούμε και ένωση περιοχών από τον πληθυσμό. Ε, σκεφτούμε πώς ε, θα κινητοποιηθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες, τα μέσα μεταφοράς κτλ. Στο σημερινό μηχανισμό δεν ξέρω αν προβλέπετε αυτό. Έχετε κοιτάξει το άρθρο 5 και το άρθρο 6 Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή λοιπόν στην υποχρέωση των κρατών μελών για να αυξήσουν τις ε, εκστρατείες ε, συνειδητοποίηση ενημέρωσης. Στα άρθρα 14 και 15 προβλέπονται κάποιες διαδικασίες που περιγράφονται με τρόπο πάρα πολύ λεπτομερή. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω καμία πρόνοια για ανάπτυξη της βοήθειας εκ των προτέρων και στην πρώτη γραμμή. Γιατί οι πρώτες αντιδράσεις και η άμεση αντίδραση είναι πιο σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν η βοήθεια ε, να χωριστεί σε δύο σκέλη. Πρώτα η κατεπίγουσα και μετά η ευρύτερη. Η δε χρηματοδότηση να έχει οροφή 630 εκατομμύρια. Εδώ αναφέρεται το ποσό 480 εκατομμυρίων από τον τίτλο 3 του προπολογισμού. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Να φύγω από την αλληλεγγύη. Ευχαριστώ κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ. Αναμένοντας ε, το σχέδιο της γνωμοδότησης. Θα κάνω κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις σε γενικές γραμμές. Η πρόταση συνολικής αύξησης του μηχανισμού για την περίοδο 2018-2020, ε, δηλαδή τα 80 εκατομμύρια, ε, με βρίσκει θετική, αν και θα πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς υλοποίησης και παρακολούθησης. Θέλω να υπογραμμίσω το εξή ε, που αναφέρεται και σε έγγραφο της Κομισιόν του Φεβρουαρίου του 2017. Το 2016 δηλώθηκε η αδυναμία ε, της συλλογική ε, ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαντήσει και στα 17 αιτήματα βοήθειας για να αντιμετωπίσει 17 πυρκαγιές. Ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν μόνο 10 και αυτό μας έδειξε ότι η Ένωση δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένη ίσως ε, για να αντιμετωπίσει καταστάσεις εκτακτής ε, ανάγκης ε, όταν εκδηλώνονται αυτές σε πολλά κράτη-μέλη πριν το χάρη πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, τρομοκρατικές επιθέσεις. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν είναι πάντοτε σε θέση να προσφέρουν βοήθεια και θα πρέπει να παρεύουμε. Σε πρακτικό επίπεδο συμφωνούμε σε δύο σημαντικά θέματα. Καταρχήν η δημιουργία ειδικών εφεδρικών πόρων, το Rescue, ε, όπου ε, δίνεται έγκριση στην Επιτροπή να έχει τα δικά της ε, επιχειρησιακά μέσα και να θετήσει μηχανισμούς για την ταχεία πρόσβαση σε αυτά τα μέσα για να, δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν ειδικέ εφεδρικές ικανότητες προκειμένου να καλυφθούν τα κενά σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, η αναθεώρηση ενός συστήματος κινήτρων για την ε, χρήση των πόρων στην Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, αυξάνοντας τα ποσοστά χρηματοδότησης και ε, το είδος ε, των, των δαπανών που γίνονται αποδεκτές. Ευχαριστώ. Έχω δύο ονόματα ακόμα. Το κύριο Ρουάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω να υλοποιηθεί το συντοματερό δυνατόν. Έχουμε ε, σεισμούς, πυρκαγιές, καλές καταστροφές που πάντοτε υπήρχαν, όμως το 2017 πήραν ε, τεράστια έκταση ε, και ε, χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Το 2017 μπορεί να θεωρηθεί μια μαύρη χρονιά. Οι κλιματικές αλλαγές έθεσαν νέες προκλήσεις, διευρύνθηκαν οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειες τους ήταν τρομερές. Η σημερινή κατάσταση πραγμάτων ε, ουσιαστικά θα παραμείνει, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, και θα έχουμε μάλλον τη νέα κανονικότητα. Βάσει αυτής της πραγματικότητας, ε, δυστυχώς, ε, θα πρέπει να συνηθίσουμε. Και όμως ακριβώς σε αυτή θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά όλοι οι λαοί, αλλά και φυσικά θα πρέπει πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη μας και τις περιφερειές μας. Για την πρόταση που έχουμε επιτάπητος, εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την ενίσχυση των εκατοτήτων ε, της Ένωσης μέσω της δημιουργίας ε, του Rescue. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια μελλοντική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική προστασία. Θα μπορούσε να αποτελεί ένα παράδειγμα πιο ισχυρής ε, ε, Ευρώπης και πιο συγκεκριμένης. Όμως το σημαντικό είναι να έχουμε τα δικά μας μέσα, ε, είτε έχουμε τα αεροσκάφη για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, είτε για μιλάμε για ένα κινητό νοσοκομείο εγώ ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδελφούς ε, για τις ε, παρεμβάσεις τους ε, και να πω ότι θα ήθελα να συνεργαστεί ο εισηγητής με την Κομισιόν και το Συμβούλιο προκειμένου το Ρέσκιο να υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Για αυτή την ενίσχυση των ικανοτήτων θέλω να υπενθυμίσω ε, ότι είναι συμπληρωματική η δύναμη αυτή, δηλαδή τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν ε, τα δικά τους μέσα, πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν ε, τη δουλειά σε εθνικό επίπεδο. Και ως μέλος αυτής της Επιτροπής ε, και ως πρώην μέλος... Ε, της ε, Επιτροπής ε, των Περιφερειών. Εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση αυτή είχα κάνει και κάποια σχόλια στην Ολομέλεια όταν συζητούσαμε τις πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Μιλάμε συγκεκριμένα ε, για σχέδια αξιολόγηση του κινδύνου που θα είναι συντονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων ε, για να προετοιμάσουμε καλύτερα τις περιφερειές μας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Μιλάμε για συνεργασία και συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης, με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στρατηγική αλλαγή με το Ταμείο Αλληλεγγύη ή με άλλη περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης διαχείρισης, παραδείγματος χάρη τα σχέδια διαχείρισης των πλημμύρων. Και επίσης ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα κονδύλια του 2020 αλλά και τα κονδύλια για την έρευνα και την κοινοτομία. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Κομισιόν και χαιρετίζω και την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Στυλιανίδη. Θα ήθελα να ευχηθώ και στον συγητή, στους κοιόδησης συγητές και στον συγητή της Επιτροπής αυτής. Ε, καλή τύχη και κάθε επιτυχία για να ολοκληρωθεί γρήγορα η εργασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σμπόγκουρτς. Ε, ευχαριστώ πολύ ε, για αυτή την έκθεση. Ε, ο εισηγητής Μπούντα και όσα είπε ο εισηγητής Μπούντα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι φυσικές καταστροφές είναι πανταχού παρούσες σε όλο τον πλανήτη και στην Ευρώπη υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος από την τρομοκρατία της, των έλεγχο των συνόρων. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτή την πρωτοβουλία. Θα πρέπει να κάνουμε σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι διάφορες καταστροφές όπως πλημμύρες, ε, ε, εργαστασιακά ατυχήματα, ε, πυρκαγιές είναι πολύ σοβαρά και είναι σημαντικό να είμαστε καλά οργανωμένοι. Για 13 χρόνια ήμουν δήμαρχος σε μια περιφέρεια 15.000 ε, ανθρώπων και θα πρέπει λοιπόν ε, να έχουμε ένα ξεκάθαρο σύστημα οργάνωσης για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο. Επίσης απαιτείται ο εθνικός συντονισμός ε, και επιπρόσθετα χρειαζόμαστε ένα συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για να μπορούν να ελοβοηθούνται όποτε προκύπτουν διάφορα προβλήματα για να μπορούν να βοηθούνται οι διάφορες χώρες και περιφέρειες αλλά και σε τοπικό επίπεδο στη γειτονιά μπορούμε να κάνουμε κάτι ε, χρειαζόμαστε καλά καταρτισμένο προσωπικό αλλά και ε, τα απαραίτητα μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Έχουμε τους επαγγελματίες, ε, το στρατό και από την άλλη έχουμε εθελοντικές δεξαμενές, έχουμε 250.000 θελοντές πυροσβέστες σε μια χώρα 2 εκατομμυρίων ε, οι οποίοι κάνουν πολλά ε, και ε, τους εκτιμούν περισσότερο από όλου στη χώρα μας διότι προστατεύουν, σώζουν τα σπίτια και τους ανθρώπους μας από καταστροφές. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα πώ να προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους σε περίπτωση που τους συμβεί κάτι και επίσης ε, πώς ε, να ε, τους προστατεύσουμε σε περίπτωση που γίνει κάποια βλάβη και να υπάρχει κάποια αποζημίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Ισχύει λοιπόν ότι αυτό το εθελοντικό προσωπικό δεν εργάζεται ε, θα πρέπει ε, γιατί σώζουν κάποιον ε, για παράδειγμα στον Πρένοβιτς το 2014 όταν ήθελαν να σώσουν ένα εργοστάσιο δεν εργάζονταν εκείνη τη στιγμή οπότε θα πρέπει να υπάρχει υποζημίωση για κάτι τέτοιο και επίσης κάτι που είπε ο κύριος Γιάκοβιτς πρέπει να είμαστε γρήγοροι στις ανταποκρίσεις μας τα πάντα θα πρέπει να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει ε, να ε, νιώθουν το σεβασμό στην κοινωνία και να ε, μπορούν να αντιδρούν γρήγορα. Θα πρέπει να αντιδρούν λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα μόλις προκύψει μια θεομηνία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό θα, να έχουμε μηχανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου αποζημιώσεις δίνονται μετά από ένα-δύο χρόνια. Θα πρέπει όλο αυτό να γίνει όμως πολύ πιο γρήγορα. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδρούν έτσι λοιπόν πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα και είναι παράδεκτο λοιπόν ε, το να μην μπορεί να ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία περιμένει ένα-δύο χρόνια για να γίνει οτιδήποτε. Κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον συνάδελφο αλλά και τους υπόλοιπους ομιλητές γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση και η βελτίωση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας είναι ένα σημαντικό στόχος. Θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο πώς λειτουργεί το Ιταλικό σύστημα σήμερα, το οποίο είναι αποκεντρωμένο αλλά πολύ αποτελεσματικό και ταυτόχρονα είναι οργανωμένο σε περιφερειακό επίπεδο και στη συνέχεια έχουμε Οργανώσει μέσω των περιφερειών ε, σε όλη την επικράτεια. Σήμερα, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν ειδικέ ομάδες οργανωμένες, συντονισμένες με αυτές των υπολείπων περιφερειών, έτσι ώστε ανάλογα με τις ανάγκες και με την περίσταση οι περιφερειακές δυνάμεις είναι μέρος αυτών όσες είναι απαραίτητες καλούνται ταχύτατα γιατί είναι οργανωμένες και έχουν όλα τα απαραίτητα είναι αυτόνομες. Ε, δεν ε, χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να εξοπλιστούν ε, κάθε φορά γιατί είναι ήδη οργανωμένες. Έτσι λοιπόν είναι αποκεντρωμένο το σύστημα γιατί οι περιφέρειες είναι αυτές που οργανώνουν και με τη σειρά τους συντονίζουν και οργανώνουν ε, τις ε, ε, δαφικές πρωτοβουλίες. Όμως μπορεί να υπάρχει και μια νοσοκομιακή μονάδα που είναι έτοιμη να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή και μέσα σε τρεις-τέσσερις ώρες, πολλές φορές και λιγότερο, σε λιγότερο χρόνο, είναι έτοιμη να ξεκινήσει αυτή η νοσοκομιακή μονάδα και είναι εντελώ αυτόνομη. Πιστεύω ότι ο μηχανισμός ε, θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή κάθε κράτος ε, βάσει της δικής του οργάνωσης να εγγυηθεί ότι θα είναι έτοιμο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να παράσχει την τάδε βοήθεια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακριβώς ε, θα αποφασίζεται παρ' το χάρη η Κροατία είναι πιο κοντά στην καταστροφή θα χρησιμοποιηθούν οι δυνάμεις της Κροατίας ή της Σλοβανία ή της Αυστρίας αναλόγως για τις ε, ανάγκες που θα προκύψουν. Το σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να είναι σχετικά γρήγορο, αλλά θα έπρεπε να μπορεί να βασιστεί στην ε, οργανωτική ικανότητα των διάφορων κρατών ε, για να μπορεί να αναλάβει δράση όπως βρίσκεται πιο κοντά πιστεύω ότι είναι ένας ε, πολύ καλός ε, ε, μηχανισμός αυτό. Θα έχουμε απλώς σε κεντρικό επίπεδο την ικανότητα να κληθεί όποιος ήδη είναι έτοιμος και να σταλεί ταχύτατα. Δηλαδή να οργανώνεται ένα σύστημα υποστήριξης των κρατών που έχουν ανάγκη σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ Ε, θα είμαι σύντομος. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη αλλά και τον εισηγητή για την υποστήριξη ε, και επίσης θα ήθελα να, να μεταφέρω όλο αυτό στον Επίτροπό μου. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανάλυση διότι δείχνει ότι η, η πρόταση ήταν αρκετά ξεκάθαρη ώστε να γίνει και κατανοητή κάποια σχόλια σχετικά με τα όσα εργαζόμαστε ε, όσον αφορά την ε, τελευταία παρέμβαση, αυτή ακριβώς είναι η ε, λογική την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Η βασική ευθύνη επαφίεται στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να παραμείνει στα κράτη-μέλη. Αρκετά μέλη ανέφεραν ότι στα κράτη-μέλη αυτό γίνεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το Rescue προτάθηκε επειδή το υπάρχον σύστημα εθελοντική της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών δεν λειτουργεί, ιδιαίτερως σε περιπτώσεις όπου τα διάφορα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα κρίσεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν διάφορες ικανότητες οι οποίες δεν υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα λοιπόν είναι ότι αν ναι, σήμερα θα θέλαμε να εκενώσουμε έναν πολίτη που πάσχει από έμπολα, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα ικανότητα. Υπήρχε στη δεξαμενή από το Λουξεμβούργο, ήταν πολύ ακριβό Όμω όμως και αφαιρέθηκε. Αυτό το οποίο προσπαθεί λοιπόν το Rescue είναι να παράσχει ένα, ε, μια δεξαμένη ε, και να χρησιμοποιείται όπου, όπου χρειάζεται ώστε να καλύπτει διάφορα κενά. Όσον αφορά τώρα την χρηματοδότηση την οποία ανέφεραν τα μέλη, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ε, σύστημα αποζημίωση τα κράτη-μέλη μας στέλνουν το λογαριασμό, το συζητάμε και στη συνέχεια το στέλνουμε την απάντηση. Δεν είναι ένα σύστημα ε, το οποίο ανταποκρίνεται σε μια υπηρεσία έκτακτων αναγκών και όσον αφορά τις ε, τροπολογίες για τον χρηματοδοτικό κανονισμό μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό με τα κράτη-μέλη. Άλλα συστήματα τα οποία είναι πιο, αποτελε... πιο ε, αποτελεσματικά όπως για παράδειγμα τα Κασκαντέρ. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε συγκεκριμένα ποσά ώρα πτήσης ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που αποφασίζουν να βοηθήσουν ένα κράτο-μέλος θα ξέρουν ποια θα είναι η χρηματοδότηση που θα λάβουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, ε, πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει ε, κεντροποίηση. Δεύτερον, ότι δεν θέλουμε να υπάρχει γραφειοκρατία. Μερικές φορές ε, βρισκόμαστε στο κέντρο ανταπόκρισης όπου έχουμε απαιτήσει από, όλες τα, από όλα τα κράτα-μέλη όπως για παράδειγμα στις φωτιές, τις δασικές πυρκαγιές στη Βόρεια Ιταλία ε, και υπάρχει καθυστέρηση λόγω εθνικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων, λόγω ε, πολιτικής. Ε, είμαστε μια υπηρεσία έκτακτων αναγκών, πρέπει να είμαστε γρήγοροι και περισσότερη γραφειοκρατία δεν θα βοηθήσει. Έτσι λοιπόν εξετάζουμε την, την όσο το δυνατόν περισσότερη απλοποίηση. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή συναντά, συζητά με κράτη-μέλη, συναντά υπουργού εξωτερικών και τονίζει ότι θα πρέπει, ότι δεν θα πρέπει να είναι πιο πολύπλοκο, δεν θα πρέπει να είναι πιο γραφειοκρατικό Κάτι ακόμα, η πολιτική ε, προστασία ε, αφορά την υποστήριξη. Η πρόληψη και η προετοιμασία είναι το βασικό κομμάτι αυτής της πρότασης. Το RescueQ δεν θα αποφέρει αποτελέσματα αν δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ετοιμότητα και η πρόληψη είναι αρκετά ικανοποιητική στα κράτη-μέλη, τουλάχιστον ε, για το μέσο κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Παρόλα αυτά όμως, τα περισσότερα χρήματα τα οποία προέρχονται προέρχονται από τον προπολογισμό της Ένωσης προέρχεται από διαρθρωτικά ταμεία ε, και ε, εφόσον αυτό δεν μπορούσε να ε, συμπεριληφθεί στο νομικό κείμενο το συμπεριλαμβάνουμε στην επικοινωνία και θα θέλαμε να σας διασφαλίσουμε ότι οι συζητήσεις με την Γενική Διεύθυνση Άγριε Κλίμα, Περιβάλλοντος έχουν ξεκινήσει σε αυτό το πλαίσιο του EMF ε, και θα πρέπει ε, να συζητήσουμε τα θέματα της πρόληψης ε, και της ετοιμότητας για να, μπορέσουμε να, για να μπορέσει να λειτουργήσει η συγκεκριμένη πρόταση. Τέλος, εγώ και οι συνάδελφοί μου στη διάθεση, βρισκόμαστε στη διάθεση του γνωμοδότη καθώς προχωράει η συγκεκριμένη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ε, εξαιρετικές παρατηρήσεις ε, που έκαναν. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά και τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν ε, για αυτά τα κανθόβη ζητήματα γιατί δυστυχώς ε, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν αυτοί οι μηχανισμοί και γι' αυτό ε, πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμούς για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε ταχύτατα. Ε, η εμπειρογνωμοσύνη των ε, συναδέλφων ε, γιατί έχουμε πολλούς συναδέλφους που ήταν δήμαρχοι και σίγουρα έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν τέτοιες καταστάσεις και σίγουρα αυτή η εμπειρία θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που να αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα μπρος για την σωτηρία ανθρώπινων ζώων. Θέλουμε όμως να έχουμε χρήσιμα αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμα, που να μας επιτρέπει να σώζουμε ανθρώπινες ζωές και να προστατεύουμε τους πολίτες. Θέλω να χαιρετήσω τη διαθεσιμότητα της Επιτροπής ε, για να χρηματοδοτήσει τις ικανότητες αυτές ε, που δεν ε, έχουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική και γρήγορη παρέμβαση. Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις τους. Thank Και εγώ σας ευχαριστώ ε, για όλη τη συζήτηση. Αναμένουμε το κείμενο της νομοδότησης. Πότε? Στις 20 Φεβρουαρίου. Στην επόμενη συνεδρίαση. Ωραία. Θα έχουμε τότε το σχέδιο εκθέσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή και προχωρούμε. of the European Investment Παρουσίαση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Δεν πρόκειται να σας αναφέρω το ιστορικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, γιατί ελπίζω να μας τα παρουσιάσουν οι ε, προσκεκλημένη. Καλωσορίζω ε, τον κύριο Χιούμπερ Κοτόνη που είναι Διευθυντής Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που θα μας παρουσιάσει το έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να απαντήσει σε ερωτήσεις που μπορεί να του κάνουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλή σας μέρα. Κυρία Μιχαήλοβα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας προσκαλέσατε σήμερα στη διακεκραμένη σας επιτροπή και σας ευχαριστώ που μας δέχεστε. Ελπίζω να συζητήσουμε, όπως είπε και η Πρόεδρος, για τα χρηματοδοτικά μέσα. Πολύ σύντομα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι επικορικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που κατέχει το 60% των μετοχών μας και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το 30% του επενδυτικού κεφαλαίου είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε γιατί ε, οι μέτοχοι ε, καθορίζουν και χαράζουν και την πολιτική μας. Τι κάνουμε εμείς κατά κύριο λόγο υποστηρίζουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, άρα προωθούμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Και αυτό το κάνουμε πάρα πολύ απλά με προϊόντα όπως είναι εγγυήσει, μικροεπενδυτικά ε, εργαλεία, κονδύλια, ε, δωρεές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα κράτη-μέλη, λοιπόν, στα 28 κράτη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Αυτό που θα ήθελα να κάνω σήμερα είναι να επικεντρωθώ στα τα ταμεία λόγω και της ε, δομής Επιτροπής σας και των ενδιαφερόντων της και πώς ε, χρηματοδοτούμε και κάτι άλλο που ακούμε πάρα πολύ συχνά στην Ευρώπη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γιατί ακούω ότι το ΕΦΣΙ δεν υποστηρίζει πάρα πολύ περιφέρειες, ε, είναι πάρα πολύ γενικό. Ε, θα ήθελα σήμερα να σας αποδείξω με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που έχω φέρει ότι ο συνδυασμός του σχεδίου Juncker, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με τα διαρθωτικά κονδύλια είναι τεράστια ε, δυνατότητα ενίσχυσης της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Για να σας δώσω μια ιδέα λοιπόν τι κάνουμε με την περιφερειακή χρηματοδότηση 1,7 δις ε, εκατομμύρια ευρώ διαχειριζόμαστε από τα διορθωτικά ταμεία και μάλιστα 1,3 δις από τον κανονισμό για την πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα επεκταθώ στη συνέχεια σε αυτό και έχουμε και εντολές για 1,4 ε, δις ε, για τα προεταξιακά μέσα. Σύνολο 3,4 με 30 εντολές. Εκτός αυτού και επιπλέον έχουμε εμπειρία ε, από κονδύλια του προϋπολογισμού 4,8 δις, 16 εντολές. Ε, είναι εδώ με κίτρινο αυτά. Και έχουμε και διαρθρωτικά ταμεία που έχουν γίνει ταμεία, μάλλον κονδύλια στα κράτη-μέλη για να ε, επενδυθούν για τον ίδιο στόχο, δηλαδή για πρωτοβουλίες των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ένα τελευταίο, ε, η πλατφόρμα MPI, τις ιδιωτικές μετοχές, αυτό το ξεκινήσαμε και είναι συμπληρωματικό για μέτρα πολιτικής που δημιουργούμε και αυτή τη στιγμή είναι στο ΕΦΣΙ, στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αποκλειστικά. Πάρα πολύ σύντομα για να δούμε πώς έχει το ΕΦΣΙ, το πρώτο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και μιλώ μόνο για τη θηρίδα που αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι ε, στην καινοτομία και την ανάπτυξη που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 5,5 δις, εκ των οποίων 2,5 είναι από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων, στο δεύτερο εύση, το δεύτερο σκέλος που εγκρίθηκε όπως γνωρίζετε γενικά επί της αρχής, θα αυξηθεί η πρικοδότηση για τις μικρομεσαίες κατά 5 δισεκατομμύρια. Τώρα ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια. Κάτι άλλο που έχει σημασία για το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι πολύ μεγάλη μόχλευση που έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να φέρουμε. 500 δις ε, νέα ε, δανειοδότηση στις μικρομεσαίες στην Ευρώπη. Ε, θα το δείτε και στην επόμενη διαφάνεια. This is uh, the achievement under, under FC1. Αυτά είναι τα επιτεύγματα του FC1. 5,5 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα έχουν δεσμευτεί 4,5 με οικονομικούς διαμεσολαβητές. Τι είναι αυτοί οι εμπορικές τράπεζες παντού στην Ευρώπη, δημόσιες τράπεζες όπως εθνικές ε, ε, τράπεζες πρόθεσης επενδύσεων, ε, διάφορα ταμεία, μικροχρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αντίστοιχα. 4,5 δις εκεί επαναλαμβάνω και 355 συναλλαγές Μέχρι στιγμής έχουμε κινητοποιήσει 82,5 ε, δισεκατομμύρια από το σύνολο 19. Δηλαδή πραγματικά 90, ε, συγγνώμη, όχι 19, ε, λειτουργεί η μόχλευση. Αυτά κάνουν οι μεσάζοντες, οι διαμεσολαβητές για να υποστηρίξουμε ε, με νέες ε, επενδύσεις, ε, μετοχές ιδιωτικού κεφαλαίου και χρηματοδότηση. Πάνω από, από 550.000 επιχειρήσεις θέλουμε να ενισχύσουμε. Έχουμε φτάσει στις 140.000 τώρα. Ε, ακούω διάφορε επικρίσεις συχνά και εδώ στην Ευρώπη, γενικά όταν ταξιδεύω ανά την Ευρώπη, ότι οι εθνικέ τράπεζε προμόθησης των επενδύσεων δεν και αναπτυξιακέ δεν συμμετέχουν. Τώρα σας ε, έχω μια ευχάριστη είδηση. Το 54% των ε, κονδυλίων προωθούνται από τράπεζες ε, επενδυτικές, κρατικές, περιφερειακές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ως μηχανισμός χρηματοδότησης στο σχέδιο Juncker ή του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θέλω τώρα να προχωρήσω λίγο παρακάτω στα διαρθρωτικά ταμεία και πάρα πολύ σύντομα ιστορικά μια αναδρομή ε, το 2007-2013. Αν κοιτάξετε το άρθρο 1083 ε, ε, υπήρξαν δύο κονδύλια του προπολογισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία. Μάλλον σε δύο σειρές γινόταν αυτή η αναφορά και από αυτή την αναφορά τι δημιουργήθηκε. Τα γνωρίζετε φαντάζομαι και ότι υπήρχε ανάγκη θα αναγνωρίσετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να μας καθοδηγήσει τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πώ από μια νομική βάση δύο σειρών θα φτιάξουμε εμεί ένα χρηματοδοτικό μέσο. Τι είχαμε δει στι προηγούμενε προγραμματικέ περιόδου. Ε, τόνους ε, εγγράφων, κατευθυντήριες γραμμές επί κατευθυντήριων γραμμών για να μας ερμηνεύουν τι θα κάναμε. Πάντως όλα αυτά ήταν καλός πιλότος και καλό σχολείο και αν δείτε ε, το 2014-2020 έχουμε τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων που είναι πολύ σημαντικός για τη δευτερογενή νομοθεσία και πολύ ειδικέ δομές το όπως λεγόμενο blending, η συνδυασμένη ε, χρηματοδότηση από το άρθρο 39 και από το Omnibus επίσης έχουμε ε, προβλέψει το συνδυασμό των διαρθωτικών ταμείων με το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Δεν θέλω να σας κουράσω με τον Τζέρεμι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλά τα κονδύλια έχουν πιάσει τόπο. 98% είναι απορρόφηση και πολύ θα ήθελα να βλέπω τέτοια απορρόφηση στα διορθωτικά ταμεία. Στον πρώτο πυλώνα έχουμε μια μόχλευση, τριπλασιάσαμε, δηλαδή ένα ευρώ στα διορθωτικά ταμεία στην αγορά έχει γίνει τρία ευρώ και κινητοποιήσαμε 240 ιδιώτες επενδυτές για να μας βοηθήσουν ε, στο πλευρό μας Παραστάτησε πολύ σημαντικό για πιλωτικό πρόγραμμα αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά επίσης θα ήθελα να φερθώ στην επόμενη διαφάνεια, στην πρωτοβουλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πολύ ειδική ε, πρόβλεψη στον κανονισμό και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να μας δίνουν εντολή για τα διορθωτικά ταμεία για να καλύπτουν τις πρώτες ζημίες όταν δίνουμε στις τράπεζες εγγυήσεις. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουμε έξι εντολές για μεγάλα ποσά στην Ισπανία ας πούμε 800 εκατομμύρια μας έχει εμπιστευτεί από τα διορθωτικά ταμεία και προβλέπεται να αυξηθεί αυτό 116 εκατομμύρια έτσι ώστε συνολικά να φτάσουμε στα 6 δις ε, δανειοδότηση σε ισπανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθ' όλη την επικράτεια της Ισπανίας. Δηλαδή από διάφορες περιφέρειες έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα, τα έχουμε συγκολήσει για να μπορέσουμε με 12 ε, συναλλαγές να ε, δανειοδοτήσουμε μικρομεσαίες. Αντίστοιχα για τη Βουλγαρία επί παραδείγματι έχουμε λάβει 102 εκατομμύρια Έχουμε υπογράψει 10 συναλλαγές. Από τα διορθωτικά ταμεία είναι αυτά τα χρήματα. Σχεδόν με όλες τις τράπεζες στη Βουλγαρία. Και ε, προβλέπεται 608 εκατομμύρια ε, να ε, δώσουμε δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ισπανία επωφελούνται, αλλά και η Φιλανδία και η Ιταλία και η Μάλτα για να ανατρέξουν στο μέλλον ε, περισσότερο σε αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύντομα, επίσης ακούω επικρίσεις ε, για τις εγγύησεις. Οι εγγύησεις αυτές δεν είναι για να βοηθούν τις τράπεζες. Τις βοηθούν, αλλά το όφελος και το κέρδος δεν θα πρέπει να μένει στην τράπεζα, αλλά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό πώς γίνεται. Πρώτον, εξασφαλίζουμε ότι οι τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν ε, τις απαιτήσει για τις εγγύησεις, τα collaterals απέναντι ε, στους δικαιούχους και έτσι αντίστοιχα θα τιμολογήσουν και τα δάνεια ε, που δίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως προς τα επιτόκια τους. Ε, το επόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρει είναι αυτή η διαφάνεια που σας δείχνει τις εντολές που έχουμε λάβει, έτσι μια ενδεικτική εικόνα, από τη Σουηδία και Εστονία μέχρι τη Τσεχική Δημοκρατία, διάφορες περιφέρειες στη Γαλλία, αλλά και την Πολωνία, Ρουμανία και Ελλάδα εκεί με επιτυχία τα έχουμε συνδυάσει αυτά με πόρους από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αν δείτε την Ελλάδα, το κάτω δεξιά παράδειγμα, πολύ πρόσφατα, 200 εκατομμύρια από τα διαστατικά ταμεία μας έχει δώσει η Ελλάδα για να τα επενδύσουμε σε διάφορα κεφάλαια αυξημένου κινδύνου ε, με τη δέουσα επιμέλεια. Έχουμε υπογράψει 7 συναλλαγές και επίκυνται και άλλες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα υποστηρίξει ορισμένα από αυτά επιλεκτικά, επιλεγμένα μάλλον με ε, την υποστήριξη με την ε, εγγύηση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό είναι σημαντικό για να συγκεντρώσει χώρους, πόρους όπως για μια χώρα όπω είναι η Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει συγχρηματοδότηση και συνδυάζοντα το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με τα κονδύλια, τα διαρθρωτικά βλέπουμε πόσο ενδιαφέρον γεννάται για τους ιδιώτες επενδυτές στην ελληνική αγορά. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός δεν αυξάνει μόνο τον όγκο, το ποσό, αλλά κινητοποιεί και ιδιώτες ε, να επενδύσουν. Το ίδιο ισχύει και για τη συνοχή. Λίγο παρακάτω. Για τα μέτρα ε, συνοχής και περιφερειακά μέτρα. Ε, χάρη στα καλά και θετικά αποτελέσματα που είχαμε από την υποστήριξη των μικρομεσαίων, έχουμε ανοιχτεί και σε νέους τομείς, ιδιαίτερα στη γεωργία. Ο Επίτροπος Χόγκαν μας έκανε μια πολύ σαφή δήλωση πριν από δύο χρόνια και είπε «Εγώ θέλω οι αγρότες να υποφελούνται από δάνεια» από δάνεια, όχι επιδοτήσεις, γιατί επιδοτήσεις είναι περιορισμένες ε, στον όγκο τους και στα ποσά που έχουμε. Θέλω να δίνετε και δάνεια στους αγρότες. Άρα είμαστε πρωτοπόροι σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και προς το παρόν έχουμε υπογράψει τρεις συναλλαγές και θα ήθελα να τονίσω και να επαναλάβω την Ιταλική περίπτωση είναι περιφερειακή χρηματοδότηση στη Γεωργία στην Ιταλία όχι εθνική και έχουμε συγκεντρώσει σε ένα σχήμα 10 ε, περιφέρειες της Ιταλίας ε, και θα έχουμε και υποστήριξη από το Μείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έτσι, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μόχλευση. Με άλλα λόγια, αντί να έχουμε μία περιφέρεια, βασιλικάτα ας πούμε, ε, που να χρησιμοποιεί ε, τα δικαιώματα που έχει μόνο στην περιφέρεια αυτή με μηδενική σχεδόν δυνατότητα μόχλευσης ε, ε, τετραπλάσια είναι εδώ αυτή τη στιγμή συνδυαστούν οι περιφέρειες πάντα με σεβασμό ότι τα κονδύλια θα είναι υπέρ των συγκεκριμένων περιφερειών έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Μαζί με το Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων ε, αποκτούμε την απαραίτητη ευελιξία για να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τετραπλάσια μόχλευση και έτσι έχουμε σχεδιάσει και το αντίστοιχο προϊόν που φαίνεται αρκετά ελκυστικό για τις τράπεζες για να συνεργαστούν μαζί μας ε, σε αυτή την υπόθεση. Έγινε μέγας λόγος για η νομοθεσία, τον κανονισμό Omnibus. Έχει σχεδόν εγκριθεί. Είναι πολλές οι καλές προθέσεις εκεί. Και θα επαναλάβουμε τη σημασία τους ε, και θα διευκολύνουμε τη χρήση. Ε, θέλω να επαναλάβω ότι η επέκταση της πρωτοβουλίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό και ευγνωμονούμε τα τρία θεσμικά όργανα που το πρότειναν και στη συνέχεια το ενέκριναν. Κομισιόν, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο είναι πολύ σημαντικό για τη δανειοδότηση. Επίσης, ε, παρατάθηκε κατά ένα χρόνο ε, η χρήση των εργαλείων ιδιωτικών μετοχών, το, equity based, δηλαδή. Επίσης, εισήχθη ε, μια, ε, ε, ένα συνδυασμό των διαρθρωτικών κονδυλίων με το Ταμείο Στρατηγικών επειδή και τα πιλωτικά προγράμματα μας έδειξαν ότι αποδίδει πάρα πολύ από τη μια να αφαιρέσουμε κάποιο βάρος από τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά για να αυξήσουμε ταυτόχρονα τη μόχλευση. Ε, ο κλάδος της γεωργίας επίσης έχει εντοπιστεί ως πάρα πολύ σημαντικός για ε, τη χρηματοδότηση τέτοιου τύπου αλλά και άλλοι τομείς όπως είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, στο μέλλον με μεγαλύτερο σύστημα ε, θα ασχοληθούμε. Τώρα δεν θέλω να σας κουράσω με τέτοιες διαφάνειες ειδικέ και τεχνικές. Βλέπουμε με τρόπο εντυπωσιακό τον αντίκτυπο του συνδυασμού της χρηματοδότησης. Εδώ αριστερά βλέπετε τη γαλάζια στήλη που είναι η νέα δανειοδότηση. Όλο αυτό το γαλάζιο εδώ είναι νέα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από διαρθρωτικά ταμεία. Αν δείτε πώς γίνεται αυτό σε συνδυασμό με το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, πολύ ψηλότερο ο αντίκτυπος. Τώρα που έχουμε λοιπόν σφιχτά δημοσιονομικά, είναι πάρα πολύ καλή συνταγή αυτή η συνδυασμή για θετικά μέτρα και για αυξημένη μόχλευση στον προπολογισμό. είναι ε, ε, καλύτερη εναλλακτική λύση για τα κράτη-μέλη που μπορούν να υποφελούνται όχι μόνο λόγω της καλύτερης μόχλευσης αλλά και επειδή το Ταμείο Στρατηγικών Επαιδήσεων έχει και ένα ιδιαίτερο τρόπο διακυβέρνησης. Και τέλος, ε, έχει και μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα στη λειτουργία του. Τώρα, ε, τι μέλη γενέστε. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Έχουμε και το Brexit και την όλη συζήτηση, αλλά και περιορισμούς δημοσιονομικούς. Οπότε, η επόμενη προγραμματική περίοδος θα είναι κάπως διαφορετική και οι πολιετής ε, πιστώσεις. Γι' αυτό θα χρειαστεί να τρέξουμε περισσότερο σε τέτοιου τύπου συνδυασμό χρηματοδότησης και χρειάζονται πολύ περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές και μόχλευση και νέος κανονισμός φυσικά θα τα αντανακλά όλα αυτά πιστεύω. Αυτό που έχει σημασία όμως και το έχω δώσει στην τέταρτη παράγραφο τα χρηματοδοτικά μέσα ε, ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ανταγωνιστικά προς τις επιδοτήσεις που έχουν και δικαίωμα ύπαρξη και συνέχεια. Τα χρηματοδοτικά μέσα αυτά θα πρέπει να είναι κομμένα και ραμμένα για συγκεκριμένε ανάγκες και έτσι να εφαρμόζονται Και θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα όταν υπάρχει δυνατότητα άντλησης νέων κεφαλαίων και να μην τρέχουμε στις ε, επιδοτήσεις. Θα τα λέει αυτά ο νέος κανονισμός. Για να γίνει όμως αυτό και τώρα δεν σας βγάλω καμιά ε, φοβερή ομιλία για το τι περιμένω ε, ε, για τις προβλέψεις μετά το 2020. Κεντρική ιδέα είναι η απλούστευση. Θα πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, τα κράτη-μέλη να έχουν δυνατότητα ταχείας αντίδρασης, ευελιξίας στα μέσα αυτά και τα νέα προϊόντα, τα χρηματοδοτικά. Και είναι ενιαίο εγχειρίδιο χρειάζεται και να είναι αξιόπιστη λογιστική έλεγχη. Παράδειγμα, όταν υλοποιήσαμε το Τζέρεμι την προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχαμε πάνω από 100 λογιστικούς ελέγχους από διαφορετικούς ελεγχθείς και κανένας δεν εμπιστευόταν το διπλανό ελεγκτή. Ε, δεν γίνεται αυτό. Στο νέο κανονισμό θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ενιαίους ελέγχους οικονομικούς, λογιστικούς ε, για να έχουμε ταχύτερη αντίδραση, μεγαλύτερο αντίκτυπο και να πιάνουν και τόπο όλα αυτά. Ευχαριστώ. Μεγαλύτερη ευελιξία επίσης. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο λόγος ε, δικό σας για σχόλια, ερωτήσεις. Ο κύριος Μοσκόρ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση έχω. Ξέρετε ότι οι άκρες βομβαξινές περιοχές ε, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι πολιτικές που έχουν ε, υλοποιηθεί έχουν αντίκτυπο σε αυτές τις πολύ εύθραστες οικονομίες και φυσικά αντιμετωπίζουν πολλές ε, δυσκολίες. Πολλές μικρές και μεσές επιχειρήσεις λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα ε, στα νούμερα, δεν τους βγαίνουν τα νούμερα. Μήπως ε, θα μπορούσατε να μου πείτε ε, ότι αν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις ξέρετε ότι τα ποσοστά μπορεί να φαίνονται ικανοποιητικά όμως οι επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρομεσαίες δεν ξέρω αν παίρνουν όλο το μερίδιο που τους ανήκει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταμάτο. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει ως αποστολή να υποστηρίξει τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις μέσω της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Γι' αυτό προϋποθέτεται για την αγορά μια σειρά καινοτόμων ε, χρηματοοικονομικών προϊόντων ε, ε, που απευθύνονται σε διάφορα ταμεία επιχειρηματικού κινδύνου, σε ιδιωτικά κεφάλαια που λειτουργούν ως ενδιάμεση. Θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε το κόστος της διαχείριση που θα μπορούσε να τροποδοθούν αυτούς τους οικονομικούς μεσάζοντες. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις ή να μας ε, πείτε ε, πώς λεπτομερώς μπορούμε να βρούμε τα ε, επιμέρους στοιχεία σε σχέση με αυτούς τους χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους με μεταξύ των χρηματοοικονομικών ε, μέσων που δεν χρησιμοποιείται πολύ ιδιαίτερα είναι η πλήθοχρηματοδότηση, το crowdfunding που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, εσείς πώς το κρίνετε, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο, ποιε είναι οι ευκαιρίες και ποια κινδύνους βλέπετε στη χρήση αυτού του μέσου. Και από όσα είδα από τις διαφάνειες που μας παρουσιάσατε, θα ήθελα να έχω ίσως ε, κάποια άλλη στιγμή περισσότερα στοιχεία για τις επιδόσεις του ΕΦΣΥ και για το ποιο είναι ο πραγματικός αντίκτυπος ε, στη ζωή των πολιτών, πόσες θέσει εργασίας έχουν ε, δημιουργηθεί και ποιες είναι οι πραγματικές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ, κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κατανοήσω την εξέλιξη των ε, χρηματοδοτικών μέσων κατόπιν ε, της ε, έναρξης λειτουργίας του ΕΦΣΙ, του Ταμείου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. και να κατανοήσω καλύτερα τα θέματα αυτά. Ξέρουμε βέβαια ότι έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά με τις Εθνικές Επενδυτικές Τράπεζες, με τη δημιουργία διαφορών πλατφόρμων που λειτουργούν ε, ως ενδιάμεσος ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ε, του ΕΦΣΙ και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες του ΕΦΣΙ και θα ήθελα να μου πείτε ποιος ήταν ο ρόλος των εθνικών τραπεζών, αν μπορούν να δοθούν κίνητρα και πώς μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα για την επόμενη φορά. Και σε δεύτερο επίπεδο θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την απλούστευση. Όταν ε, ήμουν πρόεδρος ε, του Παιδεμοντίου, ε, είχαμε και στην τύπωση της διαχείρισης των ταμείων τύπου Τζέρεμι και τελικά επειδή ήταν πολύ πολύπλοκα τα πράγματα και απαιτούνταν πολύ μεγάλες ε, προθεσμίες τα εγκαταλείψαμε όλα αυτά και ε, δημιουργήσαμε δικά μας ε, χρηματοδοτικά μέσα που μας φαίνονταν ότι λειτουργούσαν καλύτερα και γρηγορότερα. Βέβαια αυτό εν μέρη μπορεί να μας ε, ζημίωσε κιόλας, αλλά μερικές φορές έτσι γίνονται τα πράγματα. Το θέμα της απλούστευσης είναι ζωτικό ιδίως για τις ε, περιφέρειες ε, και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το θέμα πολλές φορές ε, έχει να κάνει με την επιλογή ποιων χρηματοδοτικών μέσων. Σίγουρα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί έχουν ε, και ε, ένα αποτέλεσμα, ένα φαινόμενο μόχλευσης. Φυσικά είναι καλύτερο αυτό το χρηματοδοτικό μέσο, αν θέλουμε και κάποια ε, απόδοση, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ε, τα κονδύλια αφού τα έχουμε ανακτήσει. Ε, φυσικά αναφερθήκατε στον ενιαίο έλεγχο, είναι σημαντικός αυτός, αλλά τι εννοείται με άλλα μέτρα πλούστευσης. Ευχαριστώ κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα όλη αυτή την ενημέρωση. Πάρα πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες, όσο και απαραίτητες. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, αυτό που μας χρειάζεται είναι ένα σύστημα για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτή την αλλαγή ε, και σε αυτή τη φάση του προγραμματισμού να συμμετέχουμε και εμείς και να μην βρεθούμε μας ενδιαφέρει λοιπόν και το αρχικό στάδιο του προγραμματισμού για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εδώ βλέπω ότι σε διάφορες φάσεις της προσπάθειας συμμετέχουν διάφορα κράτη-μέλη και διάφορες περιφέρειες από τα κράτη-μέλη. Αυτό πώς έγινε, εξέφρασαν εκείνες πρωτοβουλία να συμμετέχουν ή πήγατε εσείς και τις βρήκατε και τους εμπιστήσατε την προσοχή. Πώς το έμαθαν οι περιφέρειες. Και γιατί συμμετέχουν κάποια κράτη, κάποιες περιφέρειες, ενώ κάποια άλλα όχι. Είναι έλλειψη ενημέρωσης, δυνατοτήτων ή τίποτα άλλο που φταίει. Μετά, το πρόγραμμα στο οποίο αναφερθήκατε για την ε, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό πώς θα λειτουργήσει και θα, ε, πώς θα ε, τονώσει τους οικονομικούς παράγοντες και όλη την περιφέρεια για τη συνοχή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να ενισχυθεί και το ταμείο αυτό βελτιώνει την κατάσταση στην Ευρώπη. Αλλά μήπως ενταθούν οι δυσκολίες κάποιων κρατών μελών ή κάποιων περιφερειών στο εσωτερικό τους. Ε, συνήθως οι ε, επιχειρήσεις έχουν την τάση να εγκαθίστανται στα μεγάλα αστικά κέντρα ή σε ελκυστικές περιφέρειες. Μήπως υπάρχει κίνδυνος εδώ να βρεθούν σε μειονεκτική θέση κάποιες περιφέρειες. Να δημιουργήσουμε κάπου υπεραξία σε κάποια κέντρα που προσελκύουν επενδύσεις εις βάρος κάποιων άλλων περιοχών. Πώς το βλέπετε αυτό. Να μην έχουμε συγκέντρωση στις πρωτεύουσες ή σε μεγάλες πόλεις. Μπορούμε να στηρίξουμε και πιο μειονεκτούσες περιφέρειες λιγότερο αναπτυγμένες. Επιχειρήσεις από αυτές τις περιφέρειες δεν μπορεί να προτιμηθούν. Γνωρίζουμε ότι ε, περιφέρειες ε, πλήττονται από τη διαρροή και τη φυγή των εγκεφάλων. Να δείξουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ότι η Ευρώπη δεν ξεχνάει τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Ευχαριστώ. Thank you very much. These were questions from... Αυτές ήταν οι ερωτήσεις από τα ε, μέλη της Επιτροπής. Κύριε Κοτονία, αν θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. Θα προσπαθήσω να ε, απαντήσω όλες τις ερωτήσεις ε, μία-μία όσον αφορά τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ξεκίνησα, έχω ανοίξει εδώ μία διαφάνεια η οποία δείχνει μία τέτοια περιοχή στην Γαλλία, την Λογονιού ε, που είναι μία από αυτές τις ε, περιοχές όπου στην ανάλυση μας ε, έχουμε την πεποίθηση ότι η, τα ποσά των, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων είναι αρκετά μεγάλα όμως ταυτόχρονα και οι τραπέζες χρειάζονται ένα σμπρόξιμο για να υποστηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πριν ε, λάβουμε μια εντολή και πριν αποφασίσουμε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ε, εμείς αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το χάσμα το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε έχει ταυτοποιηθεί ε, ξεκάθαρα ποιο ακριβώς είναι και πώς εμείς μπορούμε να καλύψουμε το συγκεκριμένο ε, κόσμο. Ε, στη Λαγαϊουνιού, μια μικρή νήσο, είναι ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες δεν είχαν, δίσταζαν ακόμα και όσον αφορά επιχειρήσεις να δώσουν την αναγκαία ρευστότητα έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο θα κινητοποιεί τις τράπεζες να παίρνουν περισσότερο ε, ρίσκο. Αυτή θα είναι η σωστή απάντηση. Οι αριθμοί εδώ πέρα λοιπόν σας δείχνουν τι είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε ε, να ε, πετύχουμε. Έχουμε λάβει διαρθρωτικά ταμεία τα οποία ανέρχονται στα 50 εκατομμύρια Στοχεύουμε λοιπόν ε, στην ε, La Réunion ε, μαζί με την ρευστότητα παρέχουμε δηλαδή όχι μονάχα ε, παρέχουμε δηλαδή την αναγκαία ε, ρευστότητα για να μπορούν να, μπορούν να δίνονται δάνεια στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαιτείται ανάλυση της αγοράς αυτό δεν χρειάζεται στην Γαλλία οπότε είναι προσαρμοσμένο ανάλογα με κάθε κατάσταση είναι βασισμένο στο κόστος της μόχλευσης το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε την, ε, τα ποσά και στη συνέχεια θα ζητήσουμε να επαναχρησιμοποιηθούν. Προσπαθούμε ε, να ε, δημιουργήσουμε κάποια πρότυπα, όμως πρότυπα πάνω σε ένα χάσμα το οποίο θα συζητήσουμε με την διοικούσα αρχή και στη συνέχεια θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμα αναλόγως. Ε, στην ε, La Reunion ε, ελπίζουμε ότι σε μερικούς μήνες θα μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πόσες μικρομεσές βοηθήσαμε, πόσες θέσεις εργασίας διασφαλίσαμε. Το όφελος εδώ πέρα είναι ακόμα πιο σημαντικό διότι το κόστος χρηματοδότησης που παρέχουμε δεν έχει κανένα κόστος και θέλουμε λοιπόν αυτό το μηδενικό κόστος να μεταφράσουμε μεταφραστεί στο δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χρήση λοιπόν των διαρθρωτικών ταμείων ε, βοηθούν ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην πληρώνουν απολύτως ε, τίποτα. Είναι το, ε, η τράπεζα από ίδιους πόρους θα πρέπει να παρέχει. Αυτό είναι το οποίο αξιολογείται. είναι λοιπόν ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, σχετικά με το πώς βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, μεγαλύτερο βαθμό και όχι περιορισμένη στο, στην Ήπειρο αυτή καθ' αυτή. Το άλλο ερώτημα, ερώτημα από ε, την Ιταλίδα Ευρωβουλευτή. Αυτά τα εργαλεία έχουν μεγαλύτερη σημασία εκτός του να δίνουν απλά δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε ε, την Χρηματοπιστωτική Ένωση ακόμα ε, αν ε, μια ελληνική επιχείρηση πάρει ένα δάνειο κοστίζει 8% κάτι το οποίο είναι ανήκουστο αυτή την εποχή στην Γερμανία. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μπορεί να ξεπεραστεί μονάχα άμα υποστηρίξουμε καλύτερα την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και αυτό δεν θα γίνει μονάχα βασιζόμενοι στις υπάρχουσες ε, τράπεζες. Το καλύτερο παράδειγμα που μπορώ ε, να σας ε, δώσω είναι στην Βουλγαρία πριν από 7 χρόνια δώσαμε 300 εκατομμύρια στη Βουλγαρία για να υποστηρίξουμε και να αναπτύξουμε το σύστημα επισφαλών κεφαλαίων. Αν εξετάσουμε συγκεκριμένα τη Σόφια, είναι ένα από τα hot spot όσον αφορά ε, το, τα, το επισφαλές κεφάλαιο και εκεί έχουμε δώσει διαρθρωτικά ε, ταμεία, έχουμε χρησιμοποιήσει τα διαρθρωτικά ταμεία. Στόχος μας λοιπόν είναι να αναπτύξουμε νέες ε, περιοχές, νέους τομείς. Ε, μέσω του crowdfunding λοιπόν έχουμε ένα μέσο όπου, είναι ένα μέσο το οποίο υποστηρίζουμε ιδιαίτερος αυτό δεν γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε, άλλες, και σε άλλα κράτη-μέλη δεν έχουμε ακόμα την νομική βάση θα θέλαμε όμως ε, να ε, ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε τους νομοθέτες πάνω σε αυτό για να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτά τα πρότυπα αλλά και να οθήσουμε τις αγορές καλύτερα. Ναι, υποστηρίζουμε τα αναδυόμενα χρηματοπιστωτικά εργαλεία όπως είναι το crowdfunding, η μικρο μικροχρηματοδότηση και στη Γαλλία έχουμε δει αυτέ τις καλές πρακτικές ε, που τις εφαρμόζουμε και σε άλλα κράτη-μέλη. Όμως κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα και η Γερμανία ακόμα δεν έχουν έχουν ε, έναν πολύ καλό ε, νόμο όσον αφορά την μικροχρηματοδότηση. Θα πρέπει να γίνουν λοιπόν προσπάθειες που να το ξεπερνούν αυτό. Τα διαρθρωτικά ταμεία ε, υποστηρίζουν λόγω του υψηλού ρίσκου που έχουν, μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε την αγορά αναλόγως όσον αφορά τα δεδομένα του ΕΦΣΥ είναι δημόσια. Θα χαρώ να σας παράσχω ε, τα δεδομένα για να δείτε πώς ε, ε, και ποιες επιχειρήσεις έχουν υποφεληθεί από αυτά τα δάνεια. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία μπορούμε να σας δώσουμε, όμως δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή. Ε, όσον αφορά τις χώρες, ποιος ασχολείται και πότε με το κάθε θέμα, το νομοθετικό πλαίσιο είναι ε, ξεκάθαρο και όπως μάθαμε και από την τελευταία προγραμματική περίοδο ε, θα πρέπει να γίνει από την πλευρά των κρατών μελών μια εκ των υστέρων εξάντε ανάλυση και να δούμε πώς όλο αυτό έχει επηρεάσει τους διάφορους τομείς και να γίνει μια έρευνα αποτυχίας της αγοράς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, είναι επίσης ε, συμβουλευτικό και γνωρίζουμε επίσης από την, Ευρωπαϊκό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι έχουν ε, πάρα πολλές αιτήσει από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις 60 αναλύσεις τους ε, στο πλαίσιο επίσης ε, του ε, σχεδίου Juncker γίνονται αναλύσεις, με βάση αυτές γίνονται στη συνέχεια προτάσεις οι οποίες υιοθετούνται από τις εθνικές τράπεζες αλλά και από τις ευρωπαϊκές και δυστυχώς το είδαμε στην προηγούμενη περίοδο όσο φτάνουμε στο τέλος του χρονοδιογράμματος 2020 στην προκειμένη περίπτωση και τα χρήματα δεν έχουν δαπανηθεί θεσμοί όπως ο δικός μας ξαφνικά ε, πρέπει, μας ζητάνε να κάνουμε κάποιες προσπάθειες της τελευταίας στιγμής ε, και δεν είναι ε, πολύ αργά, όμως τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να αξιοποιούν το χρόνο, τις έρευνες που δεν έχουν γίνει ακόμα, αυτό ισχύει και για τα αγροτικά εργαλεία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια γρήγορη προετοιμασία, μια πρώιμη προετοιμασία. Είμαστε έτοιμοι εμείς όμως να, προετοιμαστούμε, να βοηθήσουμε οποιοδήποτε κράτο μέλος οποιαδήποτε περιφέρεια που θέλει να αναπτύξει αυτή την τεχνογνωσία και θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί μα. Ε, τώρα οι αστικές ε, σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές όλο εξαρτάται από ε, τα εργαλεία. Εμείς για παράδειγμα χρησιμοποιούμε τα εργαλεία των τραπεζών για να υποστηρίξουμε επιχειρήσεις εκτός των αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα επισφαλή κεφάλαια γενικά έχουν ε, την τάση να ζητούν ε, την καινοτομία σε αστικές περιοχές αλλά όσον αφορά τις εγγυήσεις, τα μικροδάνεια τότε στα συμβόλαιά μας με τις τράπεζες ξεκαθαρίζουμε το που θα πρέπει να πάνε τα χρήματα για παράδειγμα σε μια πρωτοβουλία στην Ισπανία στην Εστιματούρα μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Ισπανίας Έχουμε ξεκαθαρίσει το συμβόλαιό μας με τις τράπεζές μας και το τηρούν αυτό οι τράπεζες ότι οποιαδήποτε επιχείρηση από την εστιματούρα θα πρέπει Στρεμαδούρα θα πρέπει να λαμβάνει ε, την αναγκαία υποστήριξη. Εξίσου όταν κοιτάμε τις πρωτοβουλίες ε, στην Ισπανία, οι περιοχές που έχουν, έχουν συμφωνήσει ότι οι κίνδυνοι μπορούν να γίνουν ε, κοινέ. Ε, θα μας δώσετε ένα ευρώ για παράδειγμα και εμείς θα κινητοποιήσουμε 4 έως 6. Όσον αφορά όμως τις απώλειες, αυτές μπορούν να είναι κοινέ μεταξύ των περιοχών και αυτό είναι ένα από τα ωφέλη ε, διότι ενώνουμε ε, ε, περιοχές για την υποστήριξη. Τώρα το ΕΦΣΙ και η χρήση πλατφόρμων το ανέφερα σε μία από τις διαφάνειες, το ΕΦΣΙ είναι ένα εργαλείο το οποίο βασίζεται σε πλατφόρμες ή στην ιδέα της πλατφόρμες και πράγματι στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker μας ζήτησαν να δημιουργήσουμε ε, μια πλατφόρμα ε, που βλέπετε εδώ στο MOV, ε, μια πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων. Έχουμε 35 εθνικές και περιφερειακές τράπεζες σε αυτήν την ε, πλατφόρμα. Συναντόμαστε συχνά, ανταλλάσσουμε ε, βέλτιστες πρακτικές ε, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, την παρακολούθηση, ζητήματα δικαιοδοσίας και ούτω καθεξής, καλή διακυβέρνηση. με αυτόν τον τρόπο έχουμε αναπτύξει ένα προϊόν όπου ερχόμαστε ε, σε επαφή ε, με ε, εθνικά ιδρύματα προώθησης με εθνικές τράπεζες και το προσαρμόσουμε αυτό στο σχέδιο Juncker. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο αναπτύξαμε πριν από 1,5-2 χρόνια. Τρέχει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πλαίσιο συγχρηματοδότησης δεν είναι, πρόκειται για έξυπνη χρηματοδότηση διότι βοηθά τις εθνικές ε, τράπεζες να αυξήσουν ε, την τεχνογνωσία τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ε, πώς να λαμβάνουν αποφάσεις και ούτω καθεξής. Δεν αφορά λοιπόν μονάχα χρήματα απλά, αφορά έξυπνα χρήματα. Η ιδέα της πλατφόρμας λοιπόν δεν βρίσκεται μονάχα στο πλαίσιο ε, του προγράμματος ε, του σχεδίου Juncker αλλά εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή θα αναπτύξουμε λοιπόν από αυτήν την ε, πρακτική και άλλες πλατφόρμες με τράπεζες στην τράπεζα όσον αφορά τις εγγυήσεις αλλά και τις τιτροποιήσεις. Η Πιαμόντε και άλλες περιοχές το Πεδεμόντιο και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιταλίας ε, έχουν ε, λάβει υποστήριξη από τα διορθωτικά ταμεία. Έχουμε έξι βόρειες περιοχές ε, που συνεργάζονται για να υποστηρίξουν επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων στη Βόρεια Ιταλία σε μια τέτοια περιοχή δεν θα ήταν εύκολο να έχεις πρόσβαση σε τέτοια, ε, ε, σε τέτοια ποσά όμως αυτή τη στιγμή ε, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό ενώνοντας αυτές τις έξι περιφέρειες που έχουν αρκετά χρήματα ούτως ώστε να προσελκύσουν τις επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές. Είναι κάτι που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας προσωπικά διότι είναι απόδειξη σχετικά με το πώς τα διαρθρωτικά ταμεία χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό αλλά με πιο έξυπνο τρόπο από ότι στην, στον πρώτο γύρο. Είναι μια πολύ καλή απόδειξη λοιπόν σχετικά με το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να είναι τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Τώρα όσον αφορά ε, τις ε, πληρωμές υπήρξε μια διαφάνεια τα τέλη ε, σχετικά με το ότι τα τέλη είναι πολύ ακριβά στην προηγούμενη ε, περίοδο ε, στο Jeremy ε, κάναμε μία αξιολόγηση σχετικά με τα τέλη τα οποία έπρεπε να επιβάλλονται σε αυτά τα ταμεία ξεκινήσαμε με μια ε, νομοθεσία. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και αβέβαιο όμως να εφαρμοστεί αυτό και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να υπάρχει ε, νομική βεβαιότητα πάνω σε αυτό. Δεν σας ε, λέω ότι οι οδηγίες της Κομισιόν προσφέρουν νομική βεβαιότητα, όμως είναι μια βάση καλή ερμηνείας. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν, ήταν ακριβό, ε, κουραστικό, όμως για τη διαχείριση αυτών των ποσών έχουμε χρεώσει συνολικά 0,94% ε, το οποίο είναι λιγότερο από 1% και κυριολεκτικά το έργο μας ε, είναι ξεκάθαρο. Ε, σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις μπορώ να σας ενημερώσω. Γι' αυτό δεν αφορά μονάχα την δομή του προϊόντας, ε, την στρατηγική, τη συλλογή των, ποσών και στη συνέχεια να διασφαλίσουμε καθ' όλη τη διαδικασία ότι οι, οι επενδύσεις είναι ε, ασφαλείς αυτό λοιπόν είναι το ποσό ε, το οποίο έχουμε χρεώσει κατά την προηγούμενη ε, περίοδο χρηματοδότησης και τώρα με βάση το εργαλείο και τον μεσάζοντα ε, επιβάλλουμε ή όχι τέλη. Έτσι λοιπόν δεν πληρώνονται πάντοτε τέλη στις τράπεζες. Αυτό είναι λοιπόν μια δωρεάν υπηρεσία για τις τράπεζες ε, αυτό είναι ε, δύσκολο για τις τράπεζες να πρέπει να αναφέρουν και να μπορούν να αναφέρουν στα κράτη-μέλη, τα οποία με τη σειρά τους στην Κομισιόν είναι μια πολύ αναλυτική ε, αναφορά που ξεπερνά αυτό που κάνουν συνήθως στο πλαίσιο των τεχνολογικών τους συστημάτων. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια ε, Παρ' όλα αυτά όμως εμείς δεν τους χρεώνουμε, διαφέρει ε, όμως όσον αφορά τα επισφαλή κεφάλαια, εκεί ε, η αγορά βασίζεται στα τέλη ε, και αυτό δεν αφορά το να αγοράσει ο μάνατζερ την επόμενη Ferrari. Ε, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάνω σε αυτό για τα διάφορα κόστη τα οποία υπάρχουν. Υπολογίζονται με ακρίβεια ανάλογα με το μέγεθος ενός ε, τέτοιου ποσού το οποίο κυμαίνεται στο 1 με 2% του κόστους διαχείρισης θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει όλο αυτό να συμπεριληφθεί στο συνολικό ποσό και ε, το θέμα αφορά πόσο νέο ιδιωτικό κεφάλαιο ε, αυτοί οι μάνατζερ μπορούν να συλλέξουν. και αυτό αντιστοιχεί λοιπόν ε, στα όσα κερδίζουμε ακόμα και αν προέρχεται από τον δημόσιο προϋπολογισμό. Ευελπιστώ να έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Φαντάζομαι πως ναι. Ναι, και εγώ. Δώσατε πολύ λεπτομέρειες απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Με πολλές λεπτομέρειες. Και σας ευχαριστώ και προσωπικά για τα καλά παραδείγματα που δώσατε από τη Βουλγαρία γιατί έχετε δίκιο. Καταφέραμε να κάνουμε πραγματικές αλλαγές στη χώρα λόγω αυτής της στήριξης και της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων και του συνδυασμού των μέσων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η ημερησία διάταξη. Συνάδελφοι, κατόπιν έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών που έχει προγραμματιστεί για τις 12 παρατέταρτο. Αναμένω τους συντονιστές ε, να έλθουν στις 12 παρατέταρτο. Για αυτή το πρωί ολοκληρώνουμε τη συνεδρίαση εδώ.